Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε. Εγώ μιλάω τσέχικα και θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην απόψενή μας συνεδρίαση, συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανία έρευνας και ενέργειας. Ο κύριος Ρόιλ βεβαίως ε, δεν μπορεί να προεδρεύσει απόψε, θα είναι εδώ αύριο. Πριν περάσουμε στην ακρόαση για την βιομηχανική πολιτική και την ανταλλαγή απόψε με την κυρία Χέρικαρτ, υπάρχουν κάποια οργανωτικά ζητήματα. Ξεκινώντας με μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη την αυριανή. Αύριο λοιπόν. Κανονικά το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν συζήτηση με τον κύριο Ταγιάννη, τον Επιτροπό, ο οποίος όμως δεν θα είναι εδώ, οπότε αναβάλλεται η επίσκεψη του κυρίου Ταγιάννη για κάποια άλλη στιγμή. Οπότε προτείνω να ξεκινήσουμε αύριο με το σημείο 13 την γνωμοδότηση κόμη και Σόσα Βάγνερ το 14 τα οποία κανονικά θα τα βλέπαμε μετά τις ε, ψηφοφορίες. Και μετά, μετά τις ε, ψηφοφορίες θα περάσουμε μια 15 την έκθεση ΡΕΜΕΚ. Αν ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή άλλες προτάσεις, θεωρώ πως η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου θεωρώ, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ότι εγκρίνονται, οπότε τελειώσαμε με τα τυπικά και με μεγάλη μου χαρά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λάγκεν για να κάνει μια εισαγωγή στην ακροασή μας με θέμα μια νέα ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη. κύριος Λάγκεν, ο οποίος τα διευθύνει κιόλας. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σε μια φάση στην οποία οι ιδέες και η αντίληψη για μια νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική γίνονται πιο συγκεκριμένες και αυτό είναι καλό γιατί τα τελευταία χρόνια η βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη είχε παραμεληθεί και έτσι σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας ε, έχουμε κάποια εκτήματα και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα που πρέπει να ξανατεθεί, δηλαδή των ε, ανθρώπων εκείνων και των θέσεων εργασίας με προσόντα. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε μια νέα προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής και έστω να συμφωνήσουμε σε μια στρατηγική. Ξέρετε, οι ανταγωνιστέ μας παγκοσμίω ε, κινητοποιούνται. Στη Βραζιλία υπάρχει μια υπηρεσία βιομηχανικής ανάπτυξης. Ε, η Κίνα επεξεργάζεται το νέο πενταετές ε, σχέδιο, ειδικά στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε τεράστιε επενδύσεις στη βιομηχανική παραγωγή. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε. Οπότε, κυρίε και κύριοι, Έχετε δει το σχέδιο έκθεση το δικό μου. Ήδη έχω λάβει και κάποια σχόλια. Τώρα δημοσίευσε και η Κομισιόν την ανακοίνωσή της. Τότε έχουμε άλλη μια συνεισφορά για μια προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν κάτι κοινό κάτι το οποίο είναι θετικό, αλλά και κάποιες διαφορές. Να τονίσουμε λοιπόν τα κοινά. Να ε, Έχουμε δηλαδή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία και εντός της ε, Κομισιόν θα συνδυάζει τα διάφορα στοιχεία της ε, βιομηχανικής πολιτικής και θα εστιάζει σε αυτήν και θέλουμε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα Δηλαδή να μην έχουμε μόνο μία εξέταση από πλευράς βιομηχανικής πολιτικής της νομοθεσίας, αλλά να υπάρξει ίσως μία task force για να έχουμε μία εκ των προτέρων χάραξη της πολιτικής και δεύτερον να έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ του ευρωπαϊκού επίπεδου και των κρατών μελών. Γιατί αν θέλουμε να προχωρήσουμε πραγματικά πρέπει να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε καλύτερα με τα κράτη-μέλη. Και θεωρώ σωστό να θέσουμε στόχους και απαιτήσει για το πώς θα εξετάσουμε το αν έχουμε επιτύχει αυτούς τους ε, στόχους. Αυτό αναφέρεται κάπως στο τέλος στην ε, έκθεση της Κομισιόν. Εγώ θέλω να το πω πιο ξεκάθαρα. Πού θέλουμε να, να βαδίσουμε, με ποια μέσα και να δούμε ποια είναι τα μέσα και πώς ε, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα μετά. Επίσης θα πρέπει να ενσωματωθεί η βιομηχανική πολιτική γενικά σε μια μακροοικονομική πολιτική, κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής όσο πολύ, αλλά με βάση τη συζήτηση που είχαμε για το σύμφωνο σταθερότητας ε, και την οικονομική κρίση νομίζω πως είναι σαφές πως έχει μία θέση εδώ πέρα η βιομηχανική πολιτική. Και μετά να δούμε ποια μέτρα μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή το θέμα της πολιτικής καινοτομία, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, το πώς ε, θα επικεντρωθούν περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή πώς θα οδηγηθούμε σε κάποιους τομείς κλειδιά και αγορές κλειδιά στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μια προσέγγιση βεβαίως η οποία θα πρέπει έτσι να ρυθμιστεί και να χθενιστεί καλύτερα και να την δούμε συνδυασμό με την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν. Γι' αυτό έχουμε καλέσει εδώ πέρα ειδικού για να συζητήσουν αυτά τα πράγματα μαζί μας και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχουμε επιφανείς ανθρώπους για να συνεισφέρουν για το πώς θα προσεγγίσουμε με νέο τρόπο τη βιομηχανική πολιτική. Και αυτό νομίζω πώς ε, θα πρέπει να ισχύει και στο μέλλον. Εγώ το, το λέω πάρα πολύ έντονα στην έκθεσή μου, δηλαδή να αναφερθεί σε όλα τα επίπεδα η αρχή της εταιρικής σχέσης έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εμπλέκονται σε όλη τη διάρκεια της βιομηχανικής πολιτικής. Και ίσως μπορούμε να τον ισχύσουμε στην ανακοίνωση της Κομισιόν, την αρχή αυτή δηλαδή της εταιρικής σχέσης συνεργασίας. Χαίρομαι για το ότι σήμερα λοιπόν κάνουμε μια αρχή σε έναν επικοδομητικό τέτοιο διάλογο για μια νέα βιομηχανική πολιτική και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και χαίρομαι, όπως είπα, για το ότι ήδη στη σύνδεση του εθνικού με το ευρωπαϊκό επίπεδο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι έχουμε τον πρέσβη για τη βιομηχανία της Γαλλίας ο οποίος θα μας δώσει την σκοπιά του κράτους μέλους για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Κύριε Γιάκομπ, λοιπόν, έχετε τον λόγο. Κύριε Ισηγητά, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ ειλικρινά που είχατε την καλοσύνη να με, καλέσετε, να με καλέσετε σε αυτήν την συνεδρίαση διότι θεωρώ ότι το διακύβευμα της γεωργιανικής πολιτικής που πρέπει να οικοδομήσουμε βρίσκεται στο κέντρο ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και επίσης ε, γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος σας εδώ στην Επιτροπή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ελπίζω ότι θα μας βοηθήσετε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ξεπεράσουμε το πρώτο βήμα ε, που είναι ε, η ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά διαπίστωσα κύριε Σιγητά ακριβώς μέσω της ε, εκθέσεώς σας ότι η πρώτη σας εργασία ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει. Πολύ σύντομα θα ήθελα πριν ε, αναφερθώ πραγματικά στο θέμα μας ε, να διορθώσω κάτι. Ε, δηλαδή είπατε ότι, είστε, ότι είμαι πρέσβης της βιομηχανίας. νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός στο είδος μου στην Ευρώπη. γι' αυτό θα ήθελα όχι ακριβώς να διορθώσω αλλά να σας εξηγήσω ποιος είμαι και τι κάνω. Και γιατί είμαι στη θέση που ε, βρίσκομαι. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω ασχοληθεί πάντα με την βιομηχανία. Εδώ και 40 χρόνια ασχολούμαι λοιπόν με την βιομηχανία. Διεύθυνε και διευθύνω ακόμα έναν όμιλο μεσαίου μεγέθους ε, επιχειρήσεων ε, που είναι παρόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης ε, είμαι βουλευτής στην Εθνική Συνέλευση της Γαλλίας και αντιπρόεδρος ε, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βρετάνης. Τέλος, έχω διευθύνει ε, διάφορους τομείς βιομηχανικής, διάφορους τομείς της βιομηχανίας όσον αφορά δηλαδή θέσεις σε ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες κυρίως μηχανικής. Πριν από τρεις μήνες ανέλαβα τη θέση του πρέσβη της βιομηχανίας ε, και αυτό έγινε μετά από πρόταση ε, των ε, γενικών συνελεύσεων που έκανε η βιομηχανία τον προηγούμενο χρόνο και που πρότειναν λοιπόν αυτόν, αυτήν την θέση και ο κύριος Στροζή αποφάσισε να ορίσει εμένα στη θέση αυτή. Ποια είναι η θέση μου λοιπόν και τι κάνω προσπαθώ να διευκολύνω την σχέση ανάμεσα ε, στους βιομηχάνους ε, και στους πολιτικούς ε, και την κυβέρνηση στην Γαλλία. Επίσης, ξέρετε ότι στην Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια γίνεται συζήτηση όσον αφορά την βιομηχανική πολιτική και ενδεχομένως να είμαστε και λίγο πιο μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά πάντα βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και ε, ο ρόλος μου είναι να βρω την σωστή διασύνδεση ανάμεσα στο εθνικό ε, και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, ε, ρόλος μου είναι να φέρω σε επαφή τους ε, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Γαλλίας με τους αντιστοίχους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς των άλλων χωρών. Είναι ευρύ λοιπόν το φάσμα των δραστηριοτήτων μου. Εγώ δεν θέλω σήμερα να σας ε, αναφέρω την γενικότερη έποψη της Γαλλίας όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Θα ήθελα όμως να ασχοληθώ με τρία-τέσσερα σημεία τα οποία κατά την άποψή μου είναι ουσιώδους σημασίας. Πρώτο σημείο. Φυσικά η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να καταστεί μία από τις πραγματικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δέκα επόμενα χρόνια. Είναι μία βούληση η οποία έχει επιβεβαιωθεί και επομένως τώρα πρέπει να περάσουμε σε κάτι συγκεκριμένο και αποτελεσματικό. Η ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική είναι μία από τις 7 ε, σημαίνουσες πρωτοβουλίες της στρατηγικής 2020, όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολιτικοί ηθήνοντες στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν είναι απολύτως πεπισμένοι για το καλός έχει αυτής ε, της ε, πεποίθησης και πρέπει να τους πείσουμε. Γιατί πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτος λόγος, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι βιομηχανοί μας το ξέρουν ιδιαίτερα καλά γιατί το ζουν καθημερινά, δεν μπορούμε να αρκεστούμε πλέον στο να υπομένουμε ε, τις ε, ε, συνθήκες της παγκοσμιοποίησης πρέπει να κινηθούμε ενεργητικά ε, και να λειτουργήσει η παγκοσμιοποίηση με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Μονάχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να γίνουν τέτοιες κινήσεις. Η εμπορική ε, πολιτική είναι μία από τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μετά από απόφαση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως οι επιχειρήσεις μας εξαρτώνται στο εμπορικό επίπεδο από τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που πραγματεύεται η Ευρωπαϊκή, Πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω ακόμα περισσότερο λοιπόν την ανάγκη ύπαρξης κοινή ε, βιομηχανικής πολιτικής. Δεύτερος λόγος. Πολύ συχνά το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις ε, είναι όλο και πιο πολύ ευρωπαϊκό. Βεβαίως υπάρχουν οι περιβαλλοντικές ρήτρες, οι περιβαλλοντικοί κανόνες, αλλά υπάρχουν και κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό, καθώς επίσης και την εσωτερική αγορά εν γέννη. Οι αρμοδιότητες αυτές λοιπόν βρίσκονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως θα πρέπει να τις ε, παρακολουθούμε από πολύ κοντά στα πλαίσια μιας βιομηχανικής πολιτικής. Για πολλές ε, βιομηχανίες η πρώτη σημαντική αγορά είναι η ευρωπαϊκή αγορά και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στην Ευρώπη μαθαίνουν ε, να συχνοτίζονται με αγορές εκτός της εθνικής τους Αγορά. Πρέπει να μάθουν λοιπόν και να διευκολυνθούν σε αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό βήμα έτσι ώστε να ανοίξουν μετά τα φτερά τους στο παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει κι άλλο ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για το οποίο γίνεται πολλή λόγος αλλά λίγε πράξεις, λίγα έργα. Το θέμα της ε, ε, ανταγωνιστικότητας και μάλιστα της, ε, του προβλήματος που δημιουργείται στην ανταγωνιστικότητα λόγω της συναγματικής ισοτιμίας η εξέλιξη των ε, συναλλαγματικών ε, ισοτιμιών ε, μπορεί να εξουδετερώσει πλήρως όποιες προσπάθειες έχουν γίνει επί σειρά μηνών και γνωρίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Και επίσης, δεν χρειάζεται νομίζω να ε, υπενθυμίσω ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιπροσωπεύει ε, μία πρόκληση 34 δις ε, ευρώ και επομένως χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Ένα άλλο μεγάλο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να περάσω είναι ότι Βεβαίως χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει την ανακοίνωση αυτή όσον αφορά την ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική αλλά θεωρούμε ότι πολλά μπορούν ακόμα να γίνουν έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανακοίνωση αυτή και έτσι ώστε να προσπαθήσουμε ε, να την διευρύνουμε και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Για να προσανατολιστούμε προς ε, μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική, πρέπει να κινητοποιήσουμε και τις άλλες στρατηγικές πρωτοβουλίες. Μιλήσατε κύριε ε, Ισηγητά για την ε, καινοτομία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά βεβαίως πρέπει να μιλήσουμε και για το εμπόριο και για την εσωτερική αγορά υπέρ της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό πρέπει να σημαίνει ιδιαίτερος ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε στο να θεωρούμε την βιομηχανική πολιτική μονάχα μέσα από τις αρμοδιότητες της δικής σας Επιτροπής, αλλά ότι θα πρέπει να έχουμε πλέον οριζόντια προσέγγιση του ζητήματος αυτού, εάν θέλουμε μια πραγματικά ανταγωνιστική βιομηχανία. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις πολύ σημαντικές πλευρές ε, οι οποίες ε, επηρεάζονται από άλλες πρωτοβουλίες ή άλλους τομείς της Επιτροπής. Επίσης, θα πρέπει ε, οι στόχοι να εφαρμόζονται τομεακά όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Και αυτό δεν υπογραμμίζεται αρκετά στην ανακοίνωση της Επιτροπής. πρέπει οπωσδήποτε να εξευρεθούν τα μέτρα αυτά τα οποία θα επιτρέψουν την προώθηση της βιομηχανικής αριστείας σε ορισμένους ε, κυρίως τομείς ε, εχμής. Στην ε, παρούσα ε, ε, φάση της ανακοίνωσης βεβαίως ε, φαίνεται ότι λείπουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις στη δικιά σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχετε κάνει κατά αυτή την έννοια πολύ μεγάλες προσπάθειες αλλά και άλλα πράγματα μπορούν να προσθεθούν και άλλα να γίνουν δεν μπορούμε να αρκεστούμε να αναφερόμαστε μονάχα με τα λόγια σε μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια άλλων προτεραιοτήτων θα πρέπει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά την άποψή μου εάν θέλουμε να έχουμε πραγματική συνεκτικότητα και ουσία ε, στο, στο σύνολο. Η τομιακή προσέγγιση είναι ανεπαρκής, όπως έλεγα και προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάποιες συγκεκριμένες δράσεις υπέρ συγκεκριμένων τομέων, αλλά εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια πραγματικά ε, στρατηγική σκέψη όσον αφορά την κατάρτιση των ε, κατά προτεραιότητα τομέων που βεβαίως δεν θα αφορούν μονάχα τις βιομηχανίες του μέλλοντος. Βεβαίως οι βιομηχανίες του μέλλοντος, οι τομείς του μέλλοντος είναι σημαντικές, αλλά αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν μονάχα ένα μικρό ποσοστό ε, της ε, βιομηχανικής πανοπλίας της ε, Ευρώπης και είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε την ανάπτυξη των πιο παραδοσιακών τομέων της βιομηχανίας που δεν είναι ξεπερασμένη επειδή είναι πιο παραδοσιακή Εγώ γνωρίζω πολύ καλά αυτό που ονομάζουμε mechanical engineering. Και αυτή η βιομηχανία στην Ευρώπη είναι, ε, η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι ε, πρώτη στον κόσμο. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε ε, κάποια μέτρα κατά προτεραιότητα έτσι ώστε να στηρίξουμε αυτή τη βιομηχανία. Τρίτο μήνυμα οι εσωτερικέ πολιτικές της Ευρώπης ε, θα πρέπει να ευνοήσουν την ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία μα. Και αυτό βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά του θέματος. Ε, όλα στρέφονται προς την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας ε, και θα πρέπει να στρέφονται βεβαίως με σεβασμό κάποιων αρχών ε, αρχές που συζητήθηκαν επί μακρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει πάντως, και καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα, ε, να θωρακίσουμε την αντιγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας απέναντι σε ανταγωνιστές ε, οι οποίοι δυναμώνουν στην παγκόσμια αγορά γιατί ενδεχομένως δεν έχουν και τις ίδιες αρχές με εμά και τις ίδιες, τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με εμά. Εμείς ε, πρέπει να βρούμε ε, ε, στην, στην παγκοσμιοποίηση κάτι θετικό και όχι μια ε, ιδιάζουσα αρνητική κατάσταση. Επίσης, στο κείμενο της Επιτροπής ε, δεν βλέπουμε συστάσεις επί του θέματος αυτού. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την λεγόμενη κρατική πολιτική κάποιων χωρών που ασχολούνται, που καλύπτουν τον τομέα της βιομηχανίας. Αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά για την ώρα Βεβαίως ενδυνάμωση, συνέχιση ε, και εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς όπως ε, προτείνει ο κύριος Μπαρνιέ χωρίς όμως να θυγεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής ε, για βελτίωση της, των μελετών επιπτώσεων έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των ε, του αντίκτυπου που έχει η νομοθεσία ε, στις επιχειρήσεις είναι κάτι θετικό. Γιατί είναι γεγονός ότι κάποια μέτρα μπορούν να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα ε, των επιχειρήσεων. Και εγώ δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να πάρουμε τέτοιου είδους αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά την νομοθεσία πριν την εφαρμόσουμε. Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου δεν αναφέρεται καθόλου ε, εις το θέμα του ε, άνθρακα και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα το οποίο θα πρέπει να καλύψουμε, έλλειμμα της ανακοίνωσης. Όσον αφορά την έρευνα και την ε, καινοτομία, Πρόκειται εδώ για ένα θέμα το οποίο ε, έχει αποτελέσει αντικείμενο ειδική ε, ανακοίνωση και μάλιστα πρόσφατα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό ε, γιατί δεν υπάρχει λόγο σε αυτή τη φάση να το κάνω, αλλά πάντως το διακύβευμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδους σημασία. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι ε, δαπάνες ε, έρευνας σε όλο τον ε, κόσμο. Ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχει πολλαπλασιαστεί επί τέσσερα στην Κίνα τα τελευταία χρόνια και επομένως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα. Πιστεύω άλλωστε ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι κάτι πολύ θετικό και το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί μάλιστα αρκετά γρήγορα. όσον αφορά τα clusters, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της βιομηχανικής πολιτικής. Κατά την άποψή μου, ε, χρειάζεται κάτι περισσότερο από την ανακοίνωση μιας νέας στρατηγικής ε, με ορίζοντα το 2011. Πολύ σύντομα θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη μελέτη όσον αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κλάστερς. Επίσης, ε, η διευκόλυνση όσον αφορά την πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ήδη τα εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κάνει κάποιες προτάσεις. Η Γαλλία θα ήθελε κυρίως να τονίσει το γεγονός ότι θα πρέπει στην Ευρώπη να δημιουργηθεί ένα ταμείο χρηματοδότησης ε, του κεφαλαίου κινδύνου κυρίως και όχι του κεφαλαίου ε, επένδυσης γιατί αυτό το κεφάλαιο κινδύνου ε, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή από το δημόσιο. Τελευταίο σημείο κυρίες και κύριοι, η αμοιβαιότητα για την οποία πολλής λόγος γίνεται Νομίζω ότι είναι εκ των ουκάνευ της ε, ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ε, βιομηχανικής πολιτικής. Όσον αφορά τώρα την εμπορική πολιτική, έχω να πω το εξή. Αρκετά σαφώ μα λένε οι αναδυόμενε ε, οι οικονομίε, μα περιγράφουν μάλλον την στρατηγική ανάπτυξή του, που μεταξύ άλλων βασίζεται σε μη τιμολογιακή κους ε, ε, περιορισμούς. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση εδώ, γιατί η Επιτροπή άλλωστε κάνει λόγο για αυτά στην ανακοίνωσή της. Αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει όχι μόνο να αναγνωρίζουμε κάποια προβλήματα, αλλά για τα προβλήματα αυτά να κάνουμε συγκεκριμένες και πραγματιστικές προτάσεις. Πράγμα που δεν γίνεται τώρα έστω και αν ε, σήμερα ακούμε κάποιες ε, προτάσεις στην ουσία από άποψη επιχειρησιακή δεν μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία αποτελούν πλήρη σχεδόν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εκείνη θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Τέλος. Αυτές ε, οι προτάσεις θα πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη ε, στον καθορισμό των στρατηγικών ε, αναγκών της και προτεραιοτήτων της Ευρώπης. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια, το ίδιο σκεπτικό με αυτό που είχαμε 10 χρόνια πριν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι σχέσεις μας με τις ε, άλλες ε, χώρες με τις οποίες ε, θέλουμε να αναπτύξουμε εμπορικούς δεσμούς έχουν αλλάξει. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ακριβώς τι θέλουμε και να ξέρουμε πώς έχει η καινούργια κατάσταση. Τέλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε να κάνουμε μάλλον πιο αποτελεσματικά ε, τα εργαλεία εμπορικής άμυνας τα οποία έχουμε. Καλύτερη επικοινωνία με τις ε, επιχειρήσεις ε, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά. Μείωση του χρόνου εξέτασης του κάθε φακέλου που έχει υποβληθεί. Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτά ήθελα να πω κυρίες και κύριοι. Αυτά ήταν κύριε Σιγητά κάποια μηνύματα τα οποία θα ήθελα να σας μεταφέρω εξ ονόματος της Γαλλίας. Βεβαίως μπορείτε να υπολογίζετε στην ε, βοήθεια της ε, Γαλλίας για να προωθήσετε τα ζητήματα που μας απασχολούν. Μπορείτε ακόμα και προσωπικά πάνω μου να βασιστείτε ως Ευρωπαίου βιομηχάνου ε, για να συζητήσουμε μαζί και να προωθήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε Οπωσδήποτε θα συζητήσουμε αυτό το οποίο είπατε στο τέλος, δηλαδή να γίνουν πιο συγκεκριμένες ε, κάποιες προτάσεις, αλλά και πάλι σε ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο σε ένα δεύτερο ειδικό από μια νέα χώρα, νέο κράτος μέλος, που έχει πάρα πολύ μεγάλη επαφή με τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις ε, και οικογενειακές επιχειρήσεις. Χαίρομαι λοιπόν για το ότι ήρθε από τη Ρουμανία ο Μιχαήλ Μανόλιου ο οποίος είναι πρόεδρος της ε, Ένωσης ε, της Νομοσπονδίας των Ρουμανικών Επιχειρήσεων. Έχετε τον λόγο. Ονοράτα Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την ε, συνάντηση πολλοί από εσά θα διαρωτάστε για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ. Εισαγωγικά λοιπόν θα σας πω ότι είμαι Ευρωπαίος, Ρουμάνος, ε, μηχανικός, καθηγητής και ε, λόγω ενός ατυχήματος της ιστορίας προσπάθησα να οικοδομήσω τον ε, σοσιαλισμό. Και τελικά σιγά σιγά κατάλαβα ότι υπάρχει ένα θέμα management. Είμαι λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, manager σε μια επιχείρηση. Θα κάνω μια παρουσίαση PowerPoint, αλλά αν κατάλαβα καλά, ε, χωρίς PowerPoint, απλώς θα σας διανεμηθεί ένα έγγραφο. Θέλω να επικεντρωθώ σε κάποιες βασικές ιδέες και πιο συγκεκριμένα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα ποιο είναι ένα μοντέλο το οποίο οραματιζόμαστε σε σχέση με την ε, σημερινή πραγματικότητα. Δεν πιστεύω ε, στα θαύματα, αυτή είναι η δεύτερη ιδέα μου, γιατί υπάρχει ο επιστημονικός δετερμισμός και τρίτον υπάρχει η αντίληψη της ελεύθερης βούλησης. Και μια τέταρτη βασική ιδέα έχει σχέση με τον Σαντιάγκο Καλατράβα θα σας καταπλήξει ενδεχομένως αυτό το ότι αναφέρομαι στον Καλατράβα. Χτες όμως πήγα στη Λιέγη και με εντυπωσίασε κάτι. Κάτι που οι Ευρωπαίοι εν γέννη το συνδέουν με το μέλλον. Ένα σταθμός, δηλαδή που έχει σχέση με τις μεταφορές. Ο σχεδιασμός ήταν πολύ εντυπωσιακός, μια μεταλλική κατασκευή που βεβαίως μας ε, θυμίζει τη βιομηχανία. Μην ξεχνάτε ότι στηρίζω την ευρωπαϊκή βιομηχανία και πρέπει εκεί να ε, επικεντρωθούμε. Βρισκόμαστε σε μια καμπή της ιστορίας μας. Μπορούμε να ξαναγίνουμε κατακτητές όπως είχαμε υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια. Μπορούμε να διασχίσουμε τις θάλασσες, να φέρουμε τις ε, βιομηχανίες μας σε άλλες χώρες. Αλλά επανέρχομαι στο παράδοξο που εμφανίζεται. Τι συνέβη στην Ευρώπη όταν στην Κίνα παράγονται προϊόντα τα οποία πρέπει να πουληθούν στους Ευρωπαίους ανέργους. Πρέπει το παράδοξο αυτό να λυθεί. Κάποιος έλεγε κάποτε στην ιστορία ότι ό,τι χρώμα και να έχει γάτα ε, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου όταν η γάτα μπορεί να πιάσει ποντίκια. Άρα, κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για το χρώμα της γάτας, ενώ ξεχνάμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορεί η γάτα να πιάνει τα ποντίκια. Ανάμεσα στους παρισταμένους πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι που να έχει ζήσει αυτό το ιστορικό ατύχημα, δηλαδή την αναγκαστική επαναβιομηχάνηση. Στο PowerPoint αναφέρθηκα στην, υπο... στην αποβιομηχάνηση σε σχέση με τη βιομηχάνηση και την παροχή υπηρεσιών. Αυτή είναι η... ο τίτλος το ιστορικό αυτό τύχημα μου ανάγκασε για ένα διάστημα 20-30 ετών να ε, ζήσω μια σχεδιασμένη οικονομία. Δηλαδή έγινε μια προσπάθεια επιβολής έντονου εκβιομηχανισμού και συσσωρεύτηκαν πολλά προβλήματα τα οποία αναφέρονται στη διαφάνεια που έχω εδώ μπροστά μου και τα οποία θα δείτε κι εσείς ε, όταν πάρετε το χαρτί στα χέρια σας. Εν περιπτώσει, όλες αυτές οι προσπάθειες που έγιναν από, μια μεγάλη, από ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη και να μην επαναληφθούν. Κυρίως το γεγονός ότι χάθηκε ο έλεγχος ε, της οικονομικής κατάστασης. Εδώ και λίγο καιρό το ανέφερε και ο Υπουργός. Μιλάμε για την εξέλιξη οικονομικής κατάστασης σε μια χώρα που μπορεί να προκαλέσει ένα σύστημα που καλά γνωρίζουμε στην ε, ανταλλαγή και ε, κυρίως στη μαύρη οικονομία, στη μαύρη αγορά. Υπάρχουν και πενταετή προγράμματα, με αυτά δουλεύαμε στο παρελθόν. Προσπαθούσαμε να συλλάβουμε όμως μια, ένα διαφορετικό προγραμματισμό. Εδώ έτσι οι διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης, οι διάφορες περιοχές της Ευρώπης μπορούν να επικοινωνούν επί τη βάση καλών και κυρίως επαληθευμένων ε, πληροφοριών. Ιστορικά υπήρξε το 1989 και και έκτοτε ξεκίνησε ένα άλλο φαινόμενο παρόμοιο με αυτό που ε, είχε προηγηθεί. Ε, μετά την εκβιομηχάνηση υπήρχε η αποβιομηχάνηση. Περάσαμε από μια οικονομία ε, προγραμματισμένη στην οικονομία της αγοράς. Δεν καθορίζεται επακριβώς η έννοια της οικονομίας της αγοράς και θέλω να αναφερθώ σε αυτό είναι σημαντικό ο ορισμός αυτός να ξαναγραφτεί και στα έγγραφα και στη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για το μέλλον. Αυτή η νέα φάση που ξεκίνησε μετά το 1989 ε, ξεκίνησε με μια τόση ε, της οικονομίας, της παραγωγής, ε, των υπηρεσιών και μια μετάλλαξη των υπηρεσιών και φυσικά μια υποβάθμιση. Αυτό οδήγησε σε υποβάθμιση, σε πτώση του ισοζυγίου ε, συναλλαγών. Για ένα μέλος, μέρος της Ευρώπης η πτώση αυτή σήμαινε οικονομικό χάος. Ακόμα κι αν το χάος αυτό οδήγησε στη σώρευση κεφαλαίου και είχα την την ευτυχία λόγω του ιστορικού αυτού να το παρακολουθήσω και αυτό, ε, αυτό στηρίχθηκε σε σαφρές βάσεις. Οι διάφορες αυτές ε, πλευρές πρέπει να ληφθούν υπόψη στη στρατηγική και στο έγγραφο που θα συντάξουμε. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άγρια ιδιωτικοποίηση με κυριαρχή, στην κυριαρχία των γραφειοκρατών, πτώση της παραγωγικότητας εργασίας σε πολύ περιορισμένη νος management και καθόλου καθοδήγηση και δυναμισμό. Αναφέρομαι και σε κάποια ζητήματα, σε κάποια ερωτήματα που ζητούν απάντηση στην παρουσίασή μου και προσπαθώ να απαντήσω. Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες είναι να δούμε τι συμβαίνει με την ιδιωτική περιουσία. E με την πνευματική ιδιοκτησία πιθανότατα. Ποια θα είναι η ευφυής πολιτική εξομάλυνσης. Υπάρχουν τυποποίησης υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, οι πρώτες ύλε. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Πώς θα γίνει πιο πράσινη η οικονομία επίσης, επίσης και ποιος είναι ο βαθμός ε, ασφάλειας που θα πρέπει να προβλέψουμε στη διαχείριση των πρώτων υλών. Στην ανάλυση που κάνω προσπάθησα να φτιάξω ένα σχεδιάγραμμα με τα διάφορα θετικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να φτιάξουμε μια καλή πολιτική εκβιομηχάνησης και να αποφύγουμε τα αρνητικά του παρελθόντος. Και για να απλουστεύσουμε τα πράγματα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη δραστηριότητα του δημοσίου τομέα, να προωθήσουμε την ε, εθνική υπερηφάνεια και πρωτοβουλία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτά που έχουν ήδη γίνει Δηλαδή θα πρέπει να ξεπεράσουμε την βίαιη αντιπαράθεση της πυγμαχίας σε μια, ε, και με κάτι άλλο πιο ήπιο, κάτι σαν τον χορό ας πούμε, σαν μπαλέτο. Συμμετέχω σε μια μεγάλη οργάνωση εργοδοτών ε, και βεβαίως ε, ε, θεωρώ το διάλογο πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς έντονο κοινωνικό διάλογο που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό και που θα πρέπει να αποτελέσει θεμελιολίχο μιας καλύτερης πολιτικής εκβιομηχάνησης είναι το εξής. Πρέπει να έχουμε πιο τολμηρούς και δραστήριους επιχειρηματίες θα σας συγκρίνω, θα κάνω μια σύγκριση με αυτό που κάναμε στη Ρουμανία για να σας δείξω πώς μπορεί κανείς να, είναι, να δραστηριοποιηθεί περισσότερο. Κατά την παρουσίαση, στην παρουσίαση που έχω προετοιμάσει, έχω περιλάβει στοιχεία που ήδη περιείχε και το έγγραφο της Κομισιόν, την οποία ε, θα συγχαρώ, συγχαρώ τον εισηγητή. Μιλάει για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που θα λάβει υπόψη τη σαφώ τα σφάλματα του παρελθόντο. Κάτι το εξαιρετικά θετικό. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ε, δώσουμε έμφαση στην βιομηχανία χωρίς να παραμελήσουμε το τομέα των υπηρεσιών που πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είδαμε λοιπόν πως βλέπουν τα πράγματα στα νέα κράτη-μέλη και πάλι υπάρχει αυτή η προειδοποίηση να, είναι, να έχουν μια συνέπεια τα, τα μέτρα. το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Ως τρίτο μιλτή καλωσορίζω τον Ράινερ Χάμερ από ένα γερμανικό think tank, το Οικολογικό Ινστιτούτο, το οποίο πριν από λίγες ημέρες νομίζω ε, έλαβε το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό βραβείο στην Ευρώπη ως αναγνώριση της ε, πολιετούς εργασίας του στον τομέα αυτών και ελπίζω να λάβουμε κάποια συνεισφορά λοιπόν για τη συζήτησή μας. Να ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή αυτή κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. είναι ανακοίνωση αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα μεμονωμένα στοιχεία. Αναφέρω εδώ πέρα την ενσωμάτωση των διαφόρων πεδίων πολιτικής. Θα αναφερθώ λοιπόν στα σχόλια και σε εκείνα τα σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέλιξης γιατί λοιπόν αναφέρεται το έγγραφο αυτό integrated, ολοκληρωμένη και όχι αηφόρος βιομηχανική πολιτική. Αυτή είναι η σύγκρουση η οποία θεωρούμε πως υπάρχει μεταξύ ανταγωνιστικότητας και αηφορίας. Και το ερώτημα είναι πού είναι αυτή η σύγκρουση. Και αυτό λείπει εδώ πέρα από το έγγραφο αυτό και από την χάραξη της μελλοντικής ε, πορείας. Ε, εμείς ε, θεωρούμε πως θα πρέπει να τονιστεί να αναφερθεί το εάν θεωρούμε το ότι συγκρούονται αυτά τα δύο πράγματα η αηφορία και η ανάπτυξη αυτή και βεβαίως το γεγονός πως η βιομηχανική πολιτική στο παρελθόν δεν ήταν τόσο εφόρος. Επίσης νομίζω πως θα πρέπει να δούμε πού βρίσκονται οι νικητές εδώ πέρα και χαμένοι μιας βιομηχανικής πολιτικής. Κάτι το οποίο δεν θα πρέπει βεβαίω να μπερδέψουμε και να πούμε πως είναι η παλαιά, η παραδοσιακή και η νέα βιομηχανία. Οπωσδήποτε η παραδοσιακή βιομηχανία θα παραμείνει απαράλλαχτη σε πολλούς τομείς, σε κάποιους άλλους τομείς θα αλλάξει αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ποιες είναι οι επιμηχανίες εκείνες που θα χάσουν και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να υπάρξει κάτι, μια μετάβαση. Νομίζω και ο κύριος Λάγκε ανέφερε πως επιθυμητό θα ήταν η στόχη να είναι πιο σαφής, πιο ξεκάθαρη και να υπάρξει και μία παρακολούθηση που θα συνδεθεί με τους στόχους αυτούς και νομίζω και η ιδέα να συσταθεί εξ αρχής μια ομάδα παρακολούθησης και προώθησης αυτών των στόχων είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Στο έγγραφο της Κομισιόν βεβαίως αναφέρονται πολλές διαφορετικές πτυχές και με σωστό τρόπο αλλά κατά την άποψή μας λείπει μία περιγραφή του συνολικού συστήματος της αλληλεπίδρασης των διαφόρων συνθήκων του πλαισίου δηλαδή για να είναι επιτυχημένη η βιομηχανική πολιτική. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Βλέπετε πίσω μου αυτή την ωραία οθόνη και την παρουσίαση, το PowerPoint. Μια καλή τεχνολογία αλλά Δυστυχώς στο, στα ορεινά της αίθουσας δεν διακρίνεται γιατί είναι πολύ μικρή οθόνη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα του πώς μπορεί να παρουσιαστεί μια τεχνολογία αλλά ε, δεν δίνουμε βάση στο πλαίσιο. Μία λοιπόν σωστή βιομηχανική πολιτική χρειάζεται επαρκές πλαίσιο από πλευράς κράτους και κάποια άλλα στοιχεία. Äh, να στηρίξουμε την καινοτομία και να, δω, να αντιληφθούμε τη βιομηχανική πολιτική ω συστημική καινοτομία και υπάρχουν εδώ πέρα κάποια στοιχεία από τους στόχους, ε, τις ε, συνθήκες ε, και τους κανόνες αγοράς, τις υποδομές, τεχνολογίες και προϊόντα, αλλά και στην ε, συνείδηση και καταναλωτική συμπεριφορά. Και... Σημαντικό είναι η κρατική και η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική να αναπτύξει μια πιο σαφή στρατηγική και έναν οδικό χάρτη για το 2020 και 2050. Θα ήθελα επίσης να πω πως σε διάφορα επίπεδα πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή το μακροεπίπεδο πράγματι το έχουμε δει, αλλά πρέπει να δούμε το κλαδικό επίπεδο το οποίο επιγραμματικά θίγεται στο έγγραφο αυτό. Υπάρχει βεβαίως και το έγγραφο εργασίας. Τώρα το εάν θα υπάρξει στο τελικό κείμενο θα το δούμε, δηλαδή να υπάρξουν απαιτήσει σε διάφορους κλάδους και βεβαίως και διακλαδικά να το δούμε. Κάτι το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου στο έγγραφο και βεβαίως και το μικρό επίπεδο, στο επίπεδο του καταναλωτή. Από την πλευρά του πλαισίου, να σας πω να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στο Μάρμπουργκ, σε μια μικρή πανεπιστημιακή πόλη στη Γερμανία, είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε πως όλα τα νέα κτίρια θα ε, έχουν ε, ε ηλιακέ εγκαταστάσει, θερμικές ηλιακές εγκαταστάσεις, ηλιακού θερμοσύφωνε και όλοι οι ειδικοί ε, λένε πως είναι ο απλούστερο και φθηνότερος τρόπο για να προωθήσουμε την οικολογία και παρόλα αυτά αντικείμενο της συζήτησης ήταν πως έχουμε μία οικοδικτατορία το να διατάξουμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι δικτατορία, είναι βιομηχανική πολιτική. Γιατί είναι και οικονομικά λογικά, λογικό και οικολογικά λογικό και δημιουργεί και πάρα πολλές θέσεις εργασίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε μέσω αυτών των πλαισίων μπορούμε να προωθήσουμε μηχανική πολιτική και νομίζω αυτό θα πρέπει να δούμε περισσότερο. Να αναφέρω τώρα κάποιες άλλες πτυχές, τις οποίες θα ήθελα να τονίσω, τις οποίες έχω κατατάξει ε, ανάλογα με τα επίπεδα καινοτομία. Το πρώτο νομίζω το αναφέραμε δύο φορές ε, και είναι ε, σαφές νομίζω πως πρέπει να οριστούν οι στόχοι για το 2020 και όχι μόνο τους στόχους, γιατί αυτό είναι που μας διαχωρίζει από μια κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία τους στόχους να ορίσουμε, αλλά όχι τα μέσα. Τα μέσα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε, είναι σημαντικό να έχουμε στόχους δεύτερο για τις συνθήκες αγοράς Εκεί πέρα μας προξένησε έκπληξη το ότι δεν αναφέρεται καθόλου η ζήτηση εδώ πέρα. Η βιομηχανική πολιτική δεν είναι μόνο θέμα προσφοράς, αλλά χρειάζεται και μια ζήτηση. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα τις δημόσιες προμήθειες, τις οποίες δεν τις έχουμε καθόλου σκεφτεί, καθόλου. Ίσως να σκέφτηκαν πως δεν έχει σχέση με τη βιομηχανία. Αλλά οι δημόσιες προμήθειες έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην ζήτηση. Και μην ξεχνάμε πως όταν έχουμε μια μεγάλη εσωτερική αγορά όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ξεχάσουμε αυτό το τομέα είναι λάθος στις δε συνθήκες που δημιουργεί το κράτος θα ήθελα να αναφερθώ βεβαίως στους νόμους που θα πρέπει να δημιουργήσουν άγορες γιατί η βιομηχανική πολιτική και οι νέες τεχνολογίες είναι επιτυχημένες ε, όταν υιοθετηθούν και δοκιμαστούν στην εσωτερική αγορά. Δεν θα έχουμε επιτυχία μόνο αν ε, ασχολούμαστε μόνο με τις ξένες αγορές και τις εξαγωγές. Τέταρτον, στις τεχνολογίες χρειαζόμαστε βεβαίως ξεκάθαρους στόχους. Απογοητεύτηκα για το ότι στο έγγραφο αυτό αναφέρονται οι τεχνολογίες κλειδιά, αλλά οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες ε, αναφέρονται μόνο σε μία περίοδο. Δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω εδώ πέρα είναι πως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, για την επιτυχία της βιομηχανικής πολιτικής, δεν πρέπει να μειωθεί μόνο ο χρόνος προς την αγορά, διάθεση στην αγορά, αυτό το οποίο δηλαδή είναι η κλασική κατηγορία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, πως είμαστε πάρα πολύ καλοί στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά μέχρι να διατεθεί το προϊόν στην αγορά σε σύγκριση με την ε, Ιαπωνική Κινέζικη βιομηχανία είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά έχουμε ένα άλλο σοβαρότερο πρόβλημα νομίζω πως τα νέα δεν φτάνουν στον καταναλωτή. Δηλαδή έχουμε προϊόντα με μεγάλη ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά δεν αγοράζονται από τους καταναλωτές. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο για την βιομηχανία να αναπτύξει κάτι το οποίο θα έχει ζήτηση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε νέους τρόπους αν είναι να πουλήσουμε νέα και αηφόρα προϊόντα, θα πρέπει να ε, κάνουμε καμπάνιες ε, αηφορίας για τα κατάλληλα προϊόντα και όχι μόνο με μικρούς προϋπολογισμούς όπως τώρα και εθνικές καμπάνιες, αλλά με πανευρωπαϊκές εκστρατείες και μεγάλους προϋπολογισμούς και για ευρωπαϊκά προϊόντα και κορυφαία προϊόντα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με το εξής. Αυτό πάει προς την κατεύθυνση των υποδομών. Εάν δείτε τις εξελίξεις προγραμματίζονται για τα επόμενα 10-20 χρόνια, συζητάμε για τελείως νέες υποδομές παραγωγής ενέργειας νέα γενναία αυτοκινήτων ε, με νέες υποδομές, παραδείγματος χάρη ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μια νέα ανακαίνιση των κτηρίων. Οι αλλαγές αυτές τις υποδομές υπάρχουν ήδη και σε πάρα πολλές χώρες υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες κατά αυτών των αλλαγών στις υποδομές. Διαμαρτυρίες που θα καθυστερήσουν αυτές τις υποδομές δεκαετίες. Αν δεν γίνει αυτό, λοιπόν, θα είναι άσχημα τα πράγματα για την ευρωπαϊκή μηχανική πολιτική. Πρέπει λοιπόν να πούμε πως δεν είναι η κλασική οικολόγη αυτή. Αν δείτε ποιος αντιδρά σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις ενώσεις πολιτών κατά τέτοιων αποθηκευτικών αντλειών ή νέων σιδηροδρομικών γραμμών κατά μήκος του Ρήνου κτλ. Είναι πάλι οι επιχειρηματίες, δικηγόροι, marketing, είναι άλλοι δηλαδή από αυτούς που συνήθως διαμαρτύρονται. Στην οπότε πρέπει να προσέξουμε, να αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπήρχε προγραμματισμός να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός διάδρομος, έγινε και το τούνελ στην Ελβετία και στον Ρήνο θα καθυστερήσουμε πάρα πολλά χρόνια παρά το ότι είναι σαφώς, σαφές πως ε, θα αυξηθεί μεταφορά αγαθών ε, κατά 100% τα επόμενα χρόνια. Οπότε πρέπει να βρούμε νέους ε, τρόπους για αυτό, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτές τις διαφορές. Ευχαριστώ πολύ και για αυτό το οποίο είπατε, για το ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να γίνει και αποδεκτή από τους ανθρώπους και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Οι τελευταίες δύο παρουσιάσεις είναι τώρα από τους κοινωνικούς εταίρους, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι διαμορφώνουν τη βιομηχανία, από τα συνδικάτα και τους εργοδότες. Χαίρομαι για το ότι η Judith Kirten Darling είναι εδώ πέρα από την EMB, η οποία θα μας μιλήσει νομίζω από την σκοπιά της μεγαλύτερου συνδικαλιστικού οργάνου στην Ευρώπη για να μας πει τι άποψη έχουν τα συνδικάτα. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω πρώτα και καλύτερο να ευχαριστήσω την Επιτροπή που κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Μετάλλου ε, στην, ε, να διατυπώσει την άποψή της ε, για την, ε, όχι μόνο για την έκθεση της Επιτροπής, αλλά και για την ανακοίνωση της Κομισιόν. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η ακρόαση και πολύ ευπρόσδεκτη. Θέλω καταρχήν να πω ότι εκ μέρους όχι μόνο της EMF, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μια συντονισμένη προσέγγιση της, των ομοσπονδιών, των βιομηχανιών, των ορυκτών, της ενέργειας και των, του επεξεργασίας δέρματος σε σχέση με τα θέματα που ασχολείται η Κομισιόν στον τομέα της βιομηχανίας. Και εμείς ως ε, έχουμε μια άποψη ως βιομηχανικοί εργάτες για αυτά τα θέματα. Για μας το βασικό ερώτημα είναι ότι πρέπει η Ευρώπη να διατηρήσει τη φιλοδοξία της, να διατηρήσει και να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση. Η οικονομική κρίση έδειξε τη σημασία της ύπαρξης ενός βιομηχανικού ιστού στην Ευρώπη και πόσο εσφαλμένο είναι να πιστεύουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να στηρίζεται σε μια μετακίνηση προς τις υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη προσέγγιση βιομηχανία και υπηρεσίες. Και μέχρι τώρα έχουμε ακούσει πολλά, περιμένουμε όμως ε, για να δούμε και τις συγκεκριμένες προτάσεις πίσω από αυτές τις ε, εξαγγελίες. Η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική έχει προσπαθήσει να προκαταλάβει και να διαχειριστεί τις αλλαγές που συνεπάγεται η μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας προς την κατεύθυνση που θέλουμε, δηλαδή μια οικονομία που θα είναι περισσότερο βιώσιμη, που θα χρησιμοποιεί καλύτερα την ενέργεια, αλλά και που θα ε, τη χειριζόμαστε με τρόπο πιο κοινωνικά αποδεκτό και υπεύθυνο. Και αυτό φυσικά θα ε, χρειαστεί χρηματοοικονομία οικονομικά και ρυθμιστικά μέσα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην αγορά. Πρέπει να στηρίζεται σε παρέμβαση της κρατικής πολιτικής και σε ε, ξεκάθαρες ε, πολιτικές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία μας, η EMF, χαιρετίζει την νέα ανακοίνωση, όπως επίσης και την έκθεση του Bernd Lyer. Ε, πολλές καλές προτάσεις περιέχει, τις οποίες εμείς υποστηρίζουμε εδώ και καιρό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο η Ευρώπη να μην αναπτύξει μόνο μια ισχυρή ε, ε, βιομηχανική βάση αλλά και μια ένα διαφοροποιημένο βιομηχανικό ιστό που θα δώσει ε, καλές θέσεις εργασίας με μακροπρόθεσμη ορίζοντα και που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και που θεωρούμε θετικό στοιχείο στα δύο αυτά κείμενα είναι η ιδέα ότι η παραγωγή αποτελεί κομμάτι της λύσης για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες ε, αλλαγές και τις κοινωνικές ε, αλλαγές, ας πούμε, τη γύρανση της κοινωνίας ε, και τις νέες απαιτήσεις σε στον τομέα της υγείας. Η συνέχεια της υφιστάμενης διαδικασίας το οριζόντιο και στο κλαδικό χώρο είναι σημαντικές, όπως επίσης και να υπάρξουν κάποια κλαδικά, συγκεκριμένα κλαδικά προγράμματα δράσης που ε, θα απασχολήσουν ε, το ανώτατο επίπεδο ε, της Ευρώπης. Υπάρχει το θέμα της, ε, ναυπηγο, της, ναυπηγία, της ναυπηγικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, ε, του χάλιβα. Βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι πολιτικές θετικές και συγκεκριμένες που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Είναι πρόσδεκτο επίσης το γεγονός ότι και η ανακοίνωση αλλά και η έκθεση αναγνωρίζουν ότι πρέπει το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να αντιμετωπιστεί, να συμπεριληφθούν όλοι οι κλάδοι. Για μας αυτό σημαίνει μία προσέγγιση της προμηθευτικής ε, αλυσίδας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τους στρατηγικούς τομείς χωρίς να αναφερόμαστε στην εφοδιαστική αλυσίδα που τους τροφοδοτεί. Σαφώς λοιπόν είναι ευπρόσδεκτη η ολοκληρωμένη πολιτική που πρέπει να οδηγήσει σε φιλόδοξα προγράμματα επενδύσεων. Θέλουμε να ακούσουμε τι θα πει αυτή τη βδομάδα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας όσον αφορά τις ενεργειακές ε, υποδομές. Επίσης υπάρχει ε, αυτή η πρόταση για την Task Force ώστε να υπάρξει ένας μεγαλύτερος συντονισμός και μεγαλύτερη ε, συνεκτικότητα σε αυτή την προσέγγιση. Είπα λοιπόν όλα τα θετικά, όλα τα, αυτά τα οποία για μας είναι ευπρόσδεκτα, αλλά έχουμε και κάποια αιτήματα που θεωρούμε ότι αποτελούν τις αδυναμίες της, ε, της πρότασης μέχρι στιγμής. Πρώτον, και αυτό εθίγει, αλλά ε, μόνο εν συντομία. Η βιομηχανική πολιτική πρέπει να συνδέεται με τη μακροοικονομική πολιτική. Το να μιλάμε για μια φιλόδοξη ε, ε, βιομηχανική πολιτική ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μιλάμε για βασικά μέτρα λιτότητας σε εθνικό επίπεδο είναι αντίφαση, αποτελεί αντίφαση. Για να υπάρξει ένας, μια συνεκτική πολιτική πρέπει αυτή η συζήτηση να ενσωματωθεί στο ζήτημα. Και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της δημιουργίας του Eurobonds για τις επενδύσεις κλπ. Τα μέτρα λιτότητας όμως μάλλον θα αποδυναμώσουν πολλές από τις ε, επενδύσεις που πρόκειται να συζητηθούν. Αυτό είναι το μεγάλο ε, δίλημα για μας. Χρειαζόμαστε πολιτικές, δημοσιονομικές, ε, οι οποίες θα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτυξιακές και δεν θα πρέπει όχι μόνο από τη δική μας σκοπιά αλλά και συνολικά από την πλευρά των Ευρωπαίων εργαζομένων να υπάρξει ο, Ευρωπα... φόρος των συναλλαγών για να μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να προχωρήσει προς ένα πιο βιώσιμο ε, πρότυπο. Αυτό είναι το ευρύτερο μακροοικονομικό τοπίο που βλέπουμε ότι η λιτότητα αντιπαρατίθεται στην φιλοδοξία. Για μας όμως το πλέον αδύναμο σημείο του ζητήματος και γίνονται και κανένα δύο αναφορές στην έκθεση και είναι πρόσδεκτες δεν πιστεύουμε ότι κάποια ευρωπαϊκή εθνική πολιτική θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της χωρίς μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη και χωρίς την ισχυρή συμμετοχή των εργαζομένων σε κάθε σημείο της διαδικασίας. Τα θέματα της Κομισιόν έχουν ήδη τεθεί, αφορούν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα, όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομικός, ο περιβαλλοντικός, αλλά οπωσδήποτε και ο κοινωνικός πυλώνας. Και αυτό αποτελεί μέχρι στιγμής την, βιομηχανία, την, την δυναμία της βιομηχανικής πολιτικής. Υπάρχει το θέμα της ανταγωνιστικότητας που βάζει μεγάλη, ασκεί μεγάλη πίεση στις συνθήκες εργασίας. Και βεβαίω το ευρωπαϊκό επίπεδο ανταγωνιστικότητα πρέπει να στηριχθεί στην καινοτομία, στι βιομηχανικέ επενδύσει και στην ε, περιβαλλοντική και κοινωνική ποιότητα χωρίς να υπονομεύονται οι συνθήκες εργασίας, ε, η αγοραστική δύναμη που τελικά σημαίνει υπονόμευση της εσωτερικής ε, ζήτησης. Η οποία εσωτερική ζήτηση ίσως να αποτελεί και μία από τις βασικές αδυναμίες των πολιτικών που έχουν μέχρι στιγμή αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επανέρχομαι σε αυτό που ακούστηκε νωρίτερα, ότι βεβαίω πρέπει να συνδεθούν όλα αυτά με τι κρατικέ προμήθειε και να ε, μπουν, να υποστηριχθούν και να μπουν στην αγορά νέα καινοτόμα προϊόντα. Χρειαζόμαστε μια νέα κοινωνική διάσταση στι βιομηχανικέ πολιτικέ για να υπάρξει η κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τη οικονομική κρίση. Αυτό σημαίνει Χρειαζόμαστε νέα δικαιώματα στον χώρο εργασία που έχουν σχέση με την κοινωνικά υπεύθυνη αντιμετώπιση και διαχείριση τη αλλαγής. Ε, πρέπει να υπάρχει ε, η ανακοίνωση ενός νέου πλαισίου διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων για τη διαχείριση της αλλαγής. Χρειαζόμαστε ε, αξιόπιστη διαβίου ανάπτυξη και ε, εγγύηση τα ατομικά δικαιώματα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης αν θέλουμε να υπάρξει ευρωπαϊκή βιομηχανία, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής αγνοούμε εντός της ακρόασης αυτής. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι πιθανόν να εξασφαλίσουμε ότι όχι μόνο θα έχουμε βιομηχανία, αλλά και εργάτες που θα έχουν τις δεξιότητες να τις ε, λειτουργήσουν. Θέλουμε να συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες εργαζομένων ασχέτως μορφής σύμβασης και χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή ασφάλεια. Υπάρχει πρόταση για κοινωνική διάσταση αυτό το flexicurity ε, δεν είναι παρκές για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θεωρούμε ότι η, η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά έχει τεράστιες δυνατότητες για την πρόθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά οι φυστάμενες ισορροπίες εντός της ενιαίας αγοράς και η υπονόμευση των κοινωνικών δικαιωμάτων περιορίζουν τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης ολόκληρη την Ένωση και εμείς ως Ευρωπαίοι εργάτες μετάλλου είμαστε σαφώς αντίθετοι στις προσπάθειες κάποιων εργοδοτών και ε, πολυεθνικών να χρησιμοποιήσουν την παγκοσμιοποίηση και κυρίως την αναδιάρθρωση για να μπορέσουν κάποιες περιοχές, για να φέρουν σε αντιπαράθεση κάποιους κλάδους μεταξύ τους και κάποιες περιοχές μεταξύ τους. Δυστυχώς και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Αυτό δεν προέρχεται μόνο από τις ε, βιομηχανίες αλλά και τις ε, κυβερνήσεις οι οποίες χειρίζονται τις χώρες και τις φέρουν την παράθεση μεταξύ τους. Η περιφερειακή πολιτική είναι ένας βασικός ε, και σημαντικός τομέας στην ανάπτυξη ε, των θεμάτων που αφορούν την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Τέλος, χρειαζόμαστε την εμπλοκή και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην βιομηχανική, εμπορική, ε, ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σε όλα τα επίπεδα, στις, ε, στα θέματα τεχνολογίας, οικονομίας, αλλά και σε κλαθικό επίπεδο ή και σε επίπεδο επιχείρησης. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι θεμελιώδη σημασία. Ο κοινωνικός διάλογος, και αυτό με πολύ χαρά το άκουσα και από τον συνάδελφο από τη Ρουμανία, δεν είναι κάτι που πρέπει να το οργανώνουμε σε περιόδου αναδιάρθρωση, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει βάση του συστήματος ε, θεμέλιο λίθο του, του συστήματος, να υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για να εξασφαλίσουμε ότι η αναδιάρθρωση θα επιτευχθεί με τρόπο κοινωνικά διαχειρίσιμο. Πρέπει επίσης να δούμε τις διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών για να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται σωστές αξιολογήσεις και θα ε, γίνεται σωστή ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Το βασικό λοιπόν μήνυμα που θέλω να μεταφέρω, το βασικό μου μήνυμα είναι ότι η κοινωνική διάσταση της βιομηχανικής πολιτικής αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά περιορισμένη και αδύναμη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί ε, στα αιτήματά μας. Ε, και που έχουν σχέση με την πραγματική μετατροπή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, που θέλουμε να ακολουθήσει ένα πιο περισσότερο βιώσιμο ε, πρότυπο. Δύο λόγια για κάποια άλλα ζητήματα. Σαφώς ακολουθούμε την πολι, τις πολιτικές ε, ενέργειας και πρώτων υλών πολύ προσεκτικά γιατί αποτελούν ε, τομείς κλειδιά που επηρεάζουν τη βιομηχανία βεβαίως. Και οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας ενώ ε, ταυτόχρονα περιορίζονται οι επενδύσεις ε, σε ενεργειακές υποδομές είναι για μας βασικές δυσκολίες και, που θα προκύψουν στο μέλλον στη βιωσιμότητα του συστήματος μαζί όπως με άλλα ευρωπαϊκά ε, συνδικάτα πιέζουμε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχής που θα συγκεντρώνει τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, τους εκπροσώπους της υποδομής και του τομέα του εξοπλισμού και τους κοινωνικούς εταίρους για να εξασφαλίσουμε ότι τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τους ε, ευρωπαϊκούς οδικούς χάρτες. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, περιμένουμε, προσδοκούμε την πρόταση της Κομισιόν για τις πρώτες ύλες. Μία από τις αδυναμίες που ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί ε, σε στις διάφορες που γίνονται είναι η κερδοσκοπία που γίνεται στις αγορές πρώτων υλών που δημιουργεί δυσκολίες σε πολλούς κλάδους και που για μας δεν έχει ακόμα ε, αντιμετωπιστεί. Όσον αφορά την ε, πολιτική καινοτομία αναφέρθηκε αυτό, απλώς το θίξω Θέλουμε έναν ευρύτερο, πολύ ευρύτερο ορισμό της πολιτικής καινοτομίας που να περιλαμβάνει η ε, καινοτομία που να στηρίζεται στους εργαζόμενους και τη συμμετοχή τους και υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από αυτού. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα πρέπει να αναλάβει μια νέα ευθύνη να δουλέψει στην κοινωνική καινοτομία μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους. Όσον αφορά την τεχνική καινοτομία, ο στόχος του 3% εξακολουθεί να είναι ε, προσφυλής σε μας και ελπίζουμε ότι και θα αναπτυχθούν και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές για να βελτιωθεί η δυνατότητα, η δυναμικότητα των λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών και ε, να, να, ε, ε, να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες των νέων κρατών μελών. Αυτό για μας είναι σημαντικό. Τέλος, όσον αφορά την κλαδική ε, αλλαγή στη βιομηχανία. Είναι πρόσδεκτη, όπως σας είπα ήδη, η συνεχής ε, προσπάθεια να υπάρξει μια ε, ενασχόληση με τη βιομηχανική πολιτική ε, αν αντιμετωπιστεί η βιομηχανική πολιτική από τη σκοπιά της εφοδιαστικής αλυσίδας ε, και της διαχείρισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να διατηρήσει τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και, έχει, και να έχει προγράμματα για να τις διαχειριστεί και γι' αυτό είναι πρόσδεκτα τα σχέδια δράσης ε, που έχουν αναπτυχθεί για κάθε κλάδο υπάρχουν τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τα ε, για την ανακύκλωση ε, και ε, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του κόστους μακροπρόθεσμα. Οι τεχνολογίες αυτές όμως δεν θα μπορούσαν και δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τη συμμετοχή ε, των προϊόντων των παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων. Δηλαδή, οι νέες βιομηχανίες δεν θα εμφανίζονταν εκ του μηδενός αν δεν υπήρχε ο ήδη ε, υφιστάμενος βιομηχανικός ιστός. Και εξάλλου είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, προσαρμοστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές σε όλους τους κλάδους, οι οποίοι θα συνοδεύονται από επαρκή κοινωνικά μέτρα και τις συνθήκες που αφορούν την τοποθεσία για να μην υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε περιφέρειες και τόπους. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν όλα τα σημεία της ε, αλυσίδας αξιών που είναι ε, πανευρωπαϊκά. Οι εθνικές βιομηχανίες πλέον δεν υπάρχουν προσβλέπουμε στην ε, ενεργό συμμετοχή μας στη διαδικασία αυτή. Αυτό όσον αφορά την εσωτερική βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε όμως όλα αυτά τα οποία είπαμε να αναπτυχθούν και στον, στην εξωτερική ε, εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα που σημαίνει προώθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες, ε, να παίξουν ρόλο οι, οι πολυεθνικές ε, ε, και με τον τρόπο που επενδύσουν και βεβαίως να γίνονται ταχύτερες οι εκτιμήσεις των απασχολη, στην απασχόληση. Ανέφερα κάποια από τα βασικά σημεία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και των Εργατών Μετάλλου και προσβλέπουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην διατύπωση της ευρωπαϊκής πολιτικής στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την προσφορά σε βέβαιος να παίξετε έναν ε, ενεργό ρόλο και για το ότι ζητήσετε βέβαιος να γίνει κάπως πιο έντονη αυτή η θέση εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την τελευταία παρέμβαση του κυρίου Φαν Σλότεν από την σημαντική ένωση των χημικών βιομηχανιών, καθώς οι χημικές βιομηχανίες βρίσκονται σχεδόν παντού στην Ευρώπη και αποτελούν μια βιομηχανία κλειδί για την ευρωπαϊκή οικονομία. Κύριε Φανσλότεν, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Βιομηχανίας που μου δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσω την άποψη της ε, χημικής ε, βιομηχανίας ε, την ο κύκλος εργασιών είναι 450 δις ε, ε, ευρώ ε, και έχουμε περίπου, αντιπροσωπεύουμε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην κορυφή της παγκόσμιας βιομηχανίας γνωρίζετε ότι η χημική βιομηχανία ε, εφήγει, επλήγει ιδιαίτερος από την οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή όμως σιγά σιγά ξαναερχόμαστε ε, στα κανονικά μας προκρίσεως επίπεδα. Ο τομέας μας ε, όμως ε, έχει δεσμευτεί ε, να προοδεύει, να δημιουργεί θέσεις εργασίας ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Όλες οι αναλύσεις ανταγωνιστικότητας καταδεικνύουν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή θέση η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία και σιγά σιγά βρίσκουν το ρυθμό τους όλες οι περιφέρειες και ότι με, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είχαμε 32% ε, του παγκόσμιου εμπορίου. Ε, έχουμε διαρκώς βεβαίως αυξανόμενη παρουσία των αναδυόμενων οικονομιών από την ε, Ασία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός πλέον είναι παγκόσμιος. Ε, πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος δέχεται τον υφίσταται πάνω τον ανταγωνισμό από όλες τις ε, χώρες, ε, τις αναδυόμενες των αναδυόμενων ε, οικονομιών ε, και βεβαίως ε, λαμβάνονται υπόψη διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όπως είναι περιορισμοί λόγω της νέας νομοθεσίας για τις κλιματικές αλλαγές, για τις εκπομπές ρήπων κτλ. Υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες χημικές βιομηχανίες ή επιχειρήσεις στην Ευρώπη οι οποίες έχουν μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά ε, την συμμόρφωσή τους προς ε, τις ε, νομοθετικές ρυθμίσεις και επίσης αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους. Τελευταίο, αλλά σημαντικό και αυτό, η δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών και των εναλλακτικών μορφών της τροφικής αλυσίδας έτσι ώστε να γίνει πιο πράσινη η οικονομία. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την βιομηχανική ε, ε, πολιτική και στην έκθεση του κυρίου Λάγκε αναφέρονται πάρα πολλά σωστά στοιχεία όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ε, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουν την βιομηχανία τους, να κάνουν πιο ε, ε, καλή χρήση των νέων τεχνολογιών ε, και να καταφέρουν να προσαρμοστούν στη νέα οικονομία. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν τη νέα οικονομία, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να εντείνουν την συνεργασία μεταξύ των κλάστερς και να χρησιμοποιήσουν ε, στοιχεία τα οποία ήδη ε, υπάρχουν, να τα εμβαθύνουν έτσι ώστε να γίνει πιο ε, σίγουρη και σταθερή η οικονομική βάση της χημικής βιομηχανίας. Ο πρώτος λοιπόν και κυρίακος στόχος της βιομηχανίας είναι ανταγωνιστική βιομηχανία σε μια καλύτερη αηφόρο οικονομία. Ε, εμείς θέλουμε ε, να βρεθούν λύσεις απέναντι στα μεγάλα διακυβεύματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα όπως είναι ε, η πράσινη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές κτλ. Η βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να έχει παρεμβατικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορεί η βιομηχανία να ευημερεί με τον τρόπο αυτό θα έχουμε καλύτερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη χρήση ε, και ανάπτυξη των ε, πολιτικών καινοτομία. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως είναι η οικονομία, όπως είναι το εμπόριο, ε, όπως είναι το περιβάλλον. Όλες αυτές οι πολιτικές συμβάλλουν στην βελτίωση του κλίματος της βιομηχανίας. Αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η εργασία σε κλάστερς ε, και ε, η συνεργασία ε, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την δυνατότητα δημιουργίας κλάστερς καινοτομίας που ε, σχετίζονται όχι μονάχα με την χημική βιομηχανία αλλά με ολόκληρη την κατασκευαστική ε, βιομηχανία. Η χημική βιομηχανία θέτει τις βάσεις ε, για αηφόρο ανάπτυξη όχι μονάχα για την ίδια τη βιομηχανία αλλά και τις βιομηχανίες των ε, ε, συνεργατών της ε, και των πελατών της. Βρισκόμαστε επομένως στην δημιουργία ριζών που θα βοηθήσουν μέσω της καινοτομίας, θα βοηθήσουν την ανάπτυξη. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του κυρίου Λάγκε. Υπάρχουν επίσης ε, πολλά θετικά στοιχεία στην ανακοίνωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που αποτελεί μια καλή και θαραλέα αρχή. Ε, Βεβαίω, η καινοτομία θα πρέπει να ξεκινήσει και να στηριχτεί και από πολιτική και από οικονομική ε, άποψη ε, και μάλιστα να ξεκινήσει ταυτόχρονα για όλους τους τομείς. Όλες οι μελλοντικέ πολιτικές θα πρέπει να δραστηριοποιούν την αλυσίδα ε, αξιών ε, και να δημιουργεί κίνητρα και για τις ε, άλλες πολιτικές έτσι ώστε στην αγορά να φτάνουν όλο και πιο γρήγορα πραγματικά προϊόντα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την καθημερινή ζωή. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουν έρθει σε επαφή με ορισμένα στελέχη της βιομηχανίας. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Η βιομηχανία χρειάζεται όλα τα στοιχεία της έτσι ώστε να γίνει ε, σωστή, ε, να αναπτυχθεί σωστά. Ε, η χημική βιομηχανία μπορεί ε, να αποτελέσει την, ε, τον κυρίαρχο ας πούμε σε αυτήν την αλυσίδα, να είναι κατά κάποιο τρόπο value chain captain και να τεθεί επικεφαλής πολλών δράσεων που ε, μέσα από εταιρικέ σχέσει θα οδηγήσουν σε πολύ καλά αποτελέσματα. Όπως είπα και προηγουμένω, ε, η καινοτομία απαιτεί καλές, ε, μια καλή βάση δεξιοτήτων. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε δύο σημαντικές μελέτες και από την Επιτροπή αλλά και από το ΣΕΦΙΚ που κατεδεικνύει ακριβώ την ανάγκη συσχετισμού των μελλοντικών θέσεων εργασία με μια νέα βάση βάσει δεξιοτήτων. Ε, σε ολόκληρη την χημική βιομηχανία ε, γίνεται μία ε, συνεργασία έτσι ώστε να υπάρξει μία, ένας κατάλογος με τις νέες δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται η βιομηχανία για το μέλλον είναι ζωτική σημασία ε, για την βιομηχανία να έχει ε, εργαζόμενους ε, καλά προετοιμασμένους με υψηλές δεξιότητες και πολλαπλές γνώσεις το Διεθνές Έτος ε, Χημίας 2011 ε, ε, που έχει οργανωθεί υπό την αιγίδα της EUPAC και των Ηνωμένων Εθνών θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία ενδυνάμωσης του διαλόγου ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις και έτσι ώστε να καταστεί πιο ελκυστική η βιομηχανία και η χημεία γενικότερα για τους νέους ε, ταλαντούχους Ευρωπαίους. Η χημική βιομηχανία ε, ε, εξαρτάται πολύ από την δημιουργία ισχυρών κλάστες. Το ΣΕΦΙΚ πιστεύει ότι για να υπάρξει πραγματική βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, θα πρέπει να γίνεται πολλή δουλειά μέσα στα κλάστες καθώς επίσης και συνεργασία μεταξύ αυτών να δημιουργηθούν τοπικές πλατφόρμες κλάστες με ενεργή συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και των τοπικών δημοσίων αρχών εάν αυτό καταστεί απαραίτητο. Θα πρέπει επίσης ε, να υπάρξει διευρωπαϊκή συνεργασία των κλάστερς ε, χημίας και επομένως η δημιουργία τοπικών πλατφόρμων κλάστερς ε, θα πρέπει να προωθηθεί από μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα κλάστερ που, στην οποία θα αναμειχθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. καλύτερη, εξυπνότερη νομοθεσία και βελτιωμένες ε, μελέτες επιπτώσεων είναι βεβαίως πολύ ε, αξιέπαινοι οι στόχοι, αλλά αυτή τη στιγμή παραμένουν ακόμα μια ουτοπία. Η βιομηχανία πρέπει να αντιμετωπίσει μια πληθώρα ε, νομοθετικών κειμένων και ακόμα βλέπουμε πολλές ασάφειες και έλλειψη συντονισμού μεταξύ των νομικών κειμένων, ας πούμε διαφορές ανάμεσα στο RHS, στους νόμους νόμους, ε, στις οδηγίες για τα παιχνίδια, ε, στην ε, οδηγία για τα υλικά κατασκευών κτλ. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα διεθνές benchmarking ε, σε σχέση και με την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε παγκόσμια στάνταρ πιστοποίησης. Ανέφερα και την πρόσβαση στα, στις πρώτες ύλες σε καλές παγκόσμιες τιμέ. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ έτσι ώστε να έχουμε επιτυχημένη ευρωπαϊκή βιομηχανία κυρίως όσον αφορά την χημική βιομηχανία η οποία εξαρτάται τα μάλα από τις ε, ε, εισαγωγές. Ε, θα πρέπει να αρθούν μία σειρά εμποδίων ε, όπως ε, είναι τα δασμολογικά εμπόδια, τα τιμολογιακά εμπόδια κτλ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε και τα διακυβεύματα αυτά και στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Εάν η Ευρώπη πραγματικά είναι σοβαρή και θέλει πραγματικά να δημιουργήσει τις αλυσίδες αξίες, πρέπει οπωσδήποτε να άρει και τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που δημιουργούνται και απορρέουν από την κοινή γεωργική πολιτική. Οι ε, ε, υψηλή δασμοί ε, εισαγωγών όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ας πούμε η βιοεθανόλη εμποδίζει την δημιουργία σημαντικών προόδων στην ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία και βεβαίως ε, χειροτερεύουν τα πράγματα ε, μέσω της ε, χρήσης της βιομάζας που διαρκώς και μεγαλώνει λόγω των επιδοτήσεων που δίνονται από τις διάφορες χώρες. Πιστεύουμε ότι η χημική βιομηχανία μπορεί να δώσει πολλές λύσεις όσον αφορά την ανακύκλωση. Έχουμε καινοτόμια αντιμετώπιση ε, των ε, ε, διαδικασιών ανακύκλωσης. Η χημική βιομηχανία επίσης μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά την δημιουργία εναλλακτικών λύσεων σε πρώτες ύλες οι οποίες έχουν μειωθεί σε κρίσιμο επίπεδο. και βεβαίως ε, ε, συνεχίζουμε ε, την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ελάχιστη δημιουργία αποβλήτων. Για την ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία θέλουμε, έτσι ώστε να μπορέσει η, χημική, η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία να αναπτυχθεί και να γίνει ακόμα πιο δυνατή και στις περιφέρειες περιφέρειες χρειαζόμαστε μια σωστή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, η οποία δεν θα αφορά μονάχα το άνοιγμα των αγορών, αλλά και την δημιουργία, την άρση των ε, εμποδίων, αλλά και την δημιουργία αυτών των αμυντικών ε, μηχανισμών που θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα πρέπει οπωσδήποτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί και με τις χώρε χώρες ε, ΟΑΣΑ, ε, καθώς επίσης ε, και να πάρει μια υπεύθυνη θέση όσον αφορά τον τελικό γύρο της Ντόχα. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δημιουργούμε καλές γενικές συνθήκες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τα επιμέρους προβλήματα των μεμονωμένων τομέων. Οι συστάσεις της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας αποτελούν μια στρατηγική ατζέντα για θέματα, για τομείς όπως είναι η καινοτομία, ε, η ε, η πνευματική ιδιοκτησία, ε, οι νομοθετικές ρυθμίσεις, η ενέργεια, οι κλιματικές αλλαγές κλπ. Ε, ε, βρίσκουμε ότι θεωρούμε μάλλον ότι ε, αυτού του είδους ε, η συνένωση ε, τομέων βιομηχανίας που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της βρίσκουμε ότι δεν είναι η καταλληλότερη. Ο, τομέα μας, ο τομέας μας μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη απαραίτητων λύσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα οικονομία η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική ενεργειακά αλλά και θα εκπέμπει λιγότερους ρήπους εάν της δοθούν οι δυνατότητες ε, ανάπτυξης. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ολόκληρη η χημική ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία βεβαίως εξαρτάται από την πετρελαϊκή βιομηχανία σημαντικές ε, στρεβλώσεις όσον αφορά τις συνθήκες εμπορίας των πρώτων υλών, σημαντικότατες διαφορές τιμών των ε, πρώτων υλών μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, που μπορεί να υπονομεύσει το μέλλον της χημικής βιομηχανίας. Είμαστε βέβαιοι ότι εάν η Ευρώπη ε, πάρει ένα σωστό δρόμο όσον αφορά ε, την σωστή, ε, πλήρη, ολιστική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, η βιομηχανία μας θα μπορέσει να παραμείνει ηγέτης παγκόσμιος και να συνεχίσει να παίζει ρόλο όσον αφορά την συνέχεια και την ανάπτυξη της ΑΕΚ. Ευχαριστώ. Είχαμε νομίζω σαφή τοποθέτηση από την χημική βιομηχανία για ε, αυτό το οποίο ζητάτε από τη βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα λάβετε εσείς τον λόγο και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις, ε, παρατηρήσεις και τέλος ε, θα δώσω ξανά τον λόγο στους ειδικούς μας. Η κυρία Γκροστέτ ζήτησε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Αυτά που μας είπαν ε, καταδεικνύουν την ανάγκη να είμαστε φιλόδοξοι ε, για την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Φοβάμαι μην μείνουμε στα λόγια και μήπως δεν καταφέρουμε να περάσουμε στην πράξη. Αυτό ακριβώς πρέπει να προσέξουμε. Η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική να μην καταλήξει όπως η στρατηγική της Λισαβόνας από την οποία έμειναν ε, μόνο οι διακηρύξεις των προθέσεων. Ε, θέλουμε μια βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη που να είναι κάτι στο πλαίσιο της Ευρώπης του 2020 κλπ. κλπ, κλπ. Θέλουμε κάτι το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους ομιλητές για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Έχω να ρωτήσω και να σχολιάσω. Καταρχήν, πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Αν κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, πράγμα που βεβαίως επιθυμώ, πρέπει να επισέλθουμε και στις λεπτομέρειες, στη χρηματοδότηση. Υπάρχει αυτό το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Μιλήσαμε για το κεφάλαιο κινδύνου. Πρέπει να καθοριστεί τι ακριβώς θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κεφαλαίου Κινδύνου. Το αυτό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μιλήσαμε για μια ευρωπαϊκή αγορά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από καιρό την περιμένω αυτήν την Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Τι ακριβώς συμβαίνει η καταπολέμηση της ε, ε απομίμησης, ε, της ε, κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας, οι αρμοδιότητες του γραφείου, Διεθνούς Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και όλα αυτά που θα οδηγήσουν και σε κατανομή κόστους. Μια σειρά από θέματα που δεν αναφέρθηκαν υπάρχουν και οι παρεμβάσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτές χρειάζεται πολιτική θέληση, να έχουμε ενιαία φωνή. Το βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό πλέον. Άρα θα πρέπει να μιλήσουμε για πρόσβαση στις αγορές, αλλά και πάλι δεν ασχολούμαστε παρκώς με το τι εστί αμοιβαιότητα, ας πούμε, τον οικονομικό χώρο. Τι θα πει αμοιβαιότητα στην οικονομία. Γιατί όλοι μιλήσατε για τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, οι ρυθμίσεις, οι, κανονισμοί βαρύνουν τη βιομηχανία ε, και στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα της ε, το κοινωνικό. Σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα κάποια μέρα θα πούμε τι ακριβώς κάνουμε. Μήπως δεν θα πρέπει τα σύνορά μας να λάβουν υπόψη ε, το θέμα του ε, άνθρακα. Επίσης πρέπει να παρακολουθούμε, ε, να ιχνηλατούμε τα προϊόντα που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και δεν αναφερθήκαμε στη σήμανση προέλευσης που θεωρώ ότι αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό της αμοιβαιότητας. Και όταν μιλάμε για σχέση ανταγωνιστικότητας και βιομηχανίας δεν υπάρχει για μένα καμία αντιπαράθεση ανάμεσα στην ανταγωνιστική και στην βιώσιμη βιομηχανία. Πρέπει να είναι απολύτως αλληλένδετα όλα αυτά. Ε, ποια όμως είναι τα μέσα που θα δώσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη. Θα προσπαθήσουμε να αναμορφώσουμε μήπως τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να μπορούμε να εξάγουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι μια σειρά από ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε. Και βεβαίως για να μπούμε στα βαθιά θα ενισχύσουμε μια ευρωπαϊκή ή μάλλον να, θα καταφέρουμε να πετύχουμε, να δημιουργήσουμε μια πραγματική ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική χωρίς να θίξουμε τους κανόνες του ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα τολμήσουμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει η ανακοίνωση του κυρίου Ταγιάννη η οποία κατηγορείται ότι είναι ασαφής και δεν υπησέρχεται στις λεπτομέρειες. Βεβαίως διότι δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση για το τι θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική στην Κομισιόν. Υπάρχουν πολύ μεγάλη διάσταση απόψεως ανάμεσα ε, στους αρμόδιους ε, ε, επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για τον ανταγωνισμό και αυτοί οι οποίοι βεβαίως θέλουν να διατηρηθούν όλες τις εργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτηματικά τα οποία είμαστε έτοιμοι να αμφισβητήσουμε τους, κανόνες του ΠΟΕ, είμαστε έτοιμοι να αμφισβητήσουμε τους κανόνες συμφωνίες που έχουν με, συνάψει με τις τρίτες χώρες που δεν είναι πλέον αναδυόμενες, έχουν αναδυθεί. Επίσης, συμφωνούμε όπως είδαμε και πρόσφατα, καταλήξαμε να να συμπεριλάβουμε κάποιες σχετικές αναφορές σε τροποποιήσεις των συμφωνιών και εταιρικέ σχέσεις, αλλά γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνεί. Όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε ε, για να φτάσουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτούν να έχουμε αρκετή δύναμη ώστε να έχουμε βάρος απέναντι στην Κομισιόν, απέναντι στο Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με μια φωνή. Άπαξ και δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν θα έχουμε ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας και για τη δουλειά που έχετε κάνει εδώ πέρα. Ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και τους ειδικού για τις ε, ιδέες τους και τις ε, παρατηρήσεις τους οι οποίες οπωσδήποτε θα ληφθούν υπόψη. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις προς τους ε, καλεσμένους μας. Εάν ε, θεωρείτε εσείς ε, πως ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια πτυχή στην ε, βιομηχανική μας πολιτική την οποία ανέφερε η κυρία Ντάρλινγκ, δηλαδή το εργατικό δυναμικό, τους εργαζόμενους στον τομέα της βιομηχανίας που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Καθώς λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ε, κρίσης ε, οδηγηθήκαμε σε πραγματική κρίση και με τις ε, αναδιαρθρώσεις αυτές και Ξέρετε πως ε, πάρα πολλοί εργαζόμενοι με προσόντα απολύονται, κλείνουν βιομηχανίες κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το το puppy boom, το αντίθετο baby boom, δηλαδή το ότι πλέον ευνοούνται οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο δεν είναι διατραθητικό και σε πολλές βιομηχανίες, στην αεροναυτική και αλλού. Οπότε το ερώτημα τελικά είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και πως αυτό θα έπρεπε να ληφθεί στη διαμόρφωση ε, αυτής της πολιτικής. Και θα ήθελα να τονίσω και το εξής. Από τον Αμερικανικό ανταγωνισμό παρατηρούμε πως ε, η σύνδεση του στρατιωτικού με τον πολιτικό τομέα προωθεί την βιομηχανία, κάτι το οποίο δεν ισχύει τόσο πολύ στην Ευρώπη σε σύγκριση με τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή αυτή η διπλή χρήση των προϊόντων είναι κάτι το συνδυσμένο. Πάρουμε παράδειγμα την Boeing, η οποία χρησιμοποιεί τις κρατικές επιδοτήσεις που λαμβάνει για να αναπτύξει ιδιωτικά προϊόντα και μετά τα χρησιμοποιεί και στον πολιτικό τομέα. Ευχαριστώ. η Κυρία Τίκαου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ και εγώ για αυτή την έκθεση και ευχαριστώ και τους ομιλητές μας ε, οι οποίοι μίλησαν για αυτό το σημαντικό θέμα. Η βιομηχανική πολιτική βεβαίως είναι και θέμα ενεργειακής ε, αποδοτικότητας ε, που θα αποτελέσει κύριο κομμάτι της ευρωπαϊκής ατζέντα τα ευρωπαϊκά χρόνια. Και αυτό το λέω όχι μόνο γιατί θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να έχουμε ανάπτυξη και να προωθήσουμε την κοινωνική συνοχή, εάν δεν ακολουθήσει μια φιλόδοξη πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε και να σεβαστούμε το περιβάλλον και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας οι οποίες θα μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περασμένα χρόνια είχαμε αποβιομηχάνηση, μια πολιτική αποβιομηχάνησης. Δυστυχώς η παραγωγή πήγε σε χώρες που είναι φτηνότεροι και δυστυχώς και δεν υπάρχει και κοινωνική προστασία. Απλά γιατί είναι φθηνότερα τα εργατικά χέρια. Αυτό δυστυχώς οδήγησε στο ότι υπήρξε ένα χάσμα μεταξύ της καινοτομία και της έρευνας που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ένωση και έχει υπάρξει εδώ πέρα αυτό το χάσμα. Πολύ απλά έφυγε η παραγωγή και πήγε σε τρίτες χώρες. Ε, εντάξει, στιγμιαία ε, αυτό οδήγησε σε κάποια ανάπτυξη, αλλά τι εννοούμε ανάπτυξη. Ανέβηκαν οι τιμές των μετοχών των εταιριών, αλλά όχι η ίδια η αξία ε, αυτών των εταιριών, γιατί έφυγε αυτή η γνώση της παραγωγής. Οπότε από την άλλη ή από τη μία είχαμε κέρδη στις εταιρείες, από την άλλη η Ένωση έχασε σημαντικά κομμάτια της αλυσίδας από την καινοτομία μέχρι την αγορά. Και είναι σημαντικό η στρατηγική αυτή τομεί να αναγνωριστούν, να δούμε δηλαδή πού είναι ανταγωνιστική η στρατηγικη αυτη τομή να παγκοσμίω, δηλαδή αυτοκίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός, φαρμακευτικός τομέας, χημικός τομέας, αεροδιαστημική τεχνολογία. Εκεί πέρα είναι η ανταγωνιστική ένωση γιατί έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πλεόνασμα στους τομείς αυτούς, αλλά για να διατηρηθεί αυτή η ανταγωνιστικότητα και να γίνουν και άλλοι κλάδοι ανταγωνιστικοί, χρειάζεται μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική, να βρούμε δηλαδή ποιες είναι οι ικανότητες εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν σε πανεπιστημιακό επίπεδο, να δούμε πού χρειάζονται οι ειδικοί και πού θα χρειαστούν στο μέλλον και να δούμε τους τομείς κλειδιά για να έχουμε θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργία προσθέμενης αξίας έτσι ώστε στην Ευρώπη να παραμείνουν και να επανέλθουν αν θέλετε από το εξωτερικό οι ε, τομείς εκείνη της παραγωγή ε, και οι δουλειέ οι οποίε ε, έφυγαν. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πού θεωρείτε ότι πρέπει να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε θέσεις εργασίας ε, στην Ένωση, να διατηρήσουμε αυτές που έχουμε και να δημιουργήσουμε καινούργιες. Δεύτερον, ποια μέτρα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταφέρει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και παραγωγής. Γιατί φοβόμαστε πως εάν δεν γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, θα χάσουμε κάποια ικανότητα καινοτομίας και παραγωγής, γιατί δεν θα μπορούμε εδώ πέρα επί να κάνουμε ε, τα πειράματα τα οποία είναι απαραίτητα για την καινοτομία. Ευχαριστώ κύριος Σμπουτινγκόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να αναφέρω το θέμα της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής γιατί ξέρετε νηστικό αρκούδι δεν χορεύει αλλά εδώ πέρα έχει σημασία αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γκρίσχαμερ πως πρέπει να δώσουμε και θα δώσουμε πολύ δημόσιο χρήμα, αλλά δεν θα έχουμε αποτελέσματα εάν η πλευρά της ζήτησης δεν τροφοδοτηθεί από τον δημόσιο τομέα. Και είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπατε και σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος εκεί πέρα που πρέπει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Το δεύτερο που ήθελα να πω για τον τομέα της χρηματοδότησης είναι πως εγώ θα ήθελα να πω πως κυρίως όταν συζητάμε για τα δημόσια οικονομικά βλέπουμε ήδη πόσο έντονη είναι η διαμάχη μεταξύ των κρατών μελών για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και εκεί πέρα επικρατεί όχι μόνο τσιγκουνιά θα έλεγα, αλλά παραλογισμός. Και το να έχει ο καθένας ε, τους δικούς του στόχους, ε, αν θέλετε, δεν βοηθεί. Θα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς να δημιουργήσουμε το πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο στους καινοτόμους τομείς. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε τον τόνο και την έμφαση στο της, ε, σε μια βιομηχανική πολιτική που θα έχει μια λογική οριζόντια προσέγγιση και να μην καταλήξουμε σε λάθος συμπεράσματα και να οδηγηθούμε σε τομεακά μέτρα ενίσχυσης τα οποία τελικά δεν θα μπορέσουν και να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερον το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η σχέση της ανταγωνιστικότητας και της αηφορίας. Δεν θεωρώ πως είναι αντίφαση αυτό, αλλά βεβαίως αν μιλάμε για την επιβάρυνση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τις περιβαλλοντικές διατάξεις που είναι τόσο μεγάλη, ε, δεν, δεν ξέρω κι εγώ τι κατά την άποψή μου ισχύει το αντίθετο για αυτή την λεγόμενη επιβάρυνση από τις, από τις περιβαλλοντικές διατάξεις. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατά την άποψή μου θα πρέπει να λέει και ευχαριστώ στον νομοθέτη για τις περιβαλλοντικές διατάξεις γιατί όλα αυτά είναι ένα μαστίγιο καινοτομίας. Εάν αφήναμε την βιομηχανία κάθε φορά που παραπονιόταν να κάνει ό,τι θέλει, σήμερα θα ήταν λιγότερο ανταγωνιστική από ό,τι είναι de facto. Γι' αυτό θεωρώ πως ο ε, προσανατολισμός στην αηφορία είναι η βάση της βιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας και σήμερα και αύριο. Να μην το συζητάμε δηλαδή μόνο ως ένα status quo, αλλά ως κάτι το δυναμικό που θα συνεχιστεί στο μέλλον. Και μιλήσατε τώρα για τις διατάξεις, για τη φορολόγηση α, της α, ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτή είναι η βάση της οικολογικής καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Επίσης να αφαιρθώ στον κύριο Γκρίσχαμερ, δεν αντιλαμβάνομαι ε, γιατί μιλήσατε για βιομηχανίες που θα χάσουν. Γιατί ο προσανατολισμός σε μια στρατηγική που θα είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη χρήση πρώτων υλών δεν είναι κάτι το κλαδικό, είναι μια γενική στρατηγική που είναι προσβάσιμη σε όλους τους κλάδους και ε, επί της αρχής προσφέρει σε όλους την δυνατότητα να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και στο μέλλον και να ε, βγουν πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι μπήκαν σε αυτή την κατάσταση. Τέλος, ε, πάλι για τον κύριο Γκρίς Χάμπερ ε, να πω κάτι θετικό. Θεωρώ πράγματι πως δεν πρέπει να αμελήσουμε την οικονομική ενσωμάτωση το οποίο σημαίνει δύο πράγματα τουλάχιστον. Σημαίνει λογική ανάλυση συγκρούσεων που θα προκύψουν και νομίζω σωστά υπόθηκε πως η βιομηχανική πολιτική δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να την περάσουμε με το ζόρι και ε, να βρεθεί κάποιο ο οποίο θα χάσει από μία σύγκρουση, ε, νομίζω λογικό είναι να ε, προσπαθήσουμε να παίξουμε ένα προληπτικό ρόλο με τη συνεργασία και δεύτερον το γενικότερο ζήτημα τη συνείδηση τη συμπεριφοράς και τη εκπαίδευση. Θεωρώ πως και αυτό είναι ένας τομέας που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε η σημασία της ισχυρής βιομηχανίας και στο μέλλον δεν είναι κάτι το οποίο ο καθένας το αντιλαμβάνεται μόνος του, πρέπει να περάσει και στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τρεις ομιλητές θα ακούσουμε ακόμα και ε, βεβαίως μετά θα δώσω τον λόγο στους προσκεκλημένους μας να απαντήσουν. Οπότε, το γοργόν και χάριν έχει, ξέρετε. Κυρία Μέρκης. Θα σας δείξω λοιπόν ότι μπορώ να είμαι σύντομη. Σύμφωνο απόλυτα με αυτά που, με πολλά από όσα είπαν οι συνάδελφοι. Κυρίως όμως με τον τελευταίο μιλητή που είπε ότι πολύ αυστηροί περιβαλλοντικοί κανόνες προκάλεσαν καινοτομίες. Αυτός είναι ένας από τους δρόμους που ανοίγονται μπροστά μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και τους συναδέλφους για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους. Με τα χαράς άκουσα πολύ να χρησιμοποιούνται οι όροι πρώτες ύλε και καινοτομία στη συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική. Τα θεωρώ αλληλένδετα τα ζητήματα αυτά. Όμως δεν άκουσα τον όρο ενιαία αγορά. Το ζήτημα δηλαδή του πώς μπορεί η ενιαία αγορά να οδηγήσει σε μια βιομηχανική πολιτική. Καινοτομία και ενιαία αγορά. Πώς θα προσφέρουμε δε στη βιομηχανία μας τις πρώτε και θα έχουμε επαρκείς εναλλακτικέ λύσεις. Όλα αυτά έχουν άμεση, άρρηκτη σχέση μεταξύ τους. Ξέρετε πόσο με ενδιαφέρει το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας για τον τρόπο με τον οποίο τις, να συνδυάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα πολιτικής ε, ίσως ήταν στο πρώτο κομμάτι και δεν το άκουσα, το θέμα της ε, συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανική πολιτική. Γιατί η βιομηχανία δεν είναι μόνο τα μεγάλα συγκροτήματα, αλλά και οι μικρές μονάδες. Και μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο η τυποποίηση η παγκόσμια αλλά και η ευρωπαϊκή θα σας βοηθήσει στον τομέα της καινοτομίας αλλά και στη βιομηχανική πολιτική. Κύριε Βαν Σλότεν, σας άκουσα να λέτε ότι η Κομισιόν ακούει μόνο έναν ή δύο από τους εμπλεκόμενους. Δεν σας κατάλαβα καλά. Α, γιατί... Ε, ίσως Είπατε ότι δεν παρακολούθησαν όλους τους εμπλεκόμενους. Α, δεν σας κατάλαβα καλά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η Κομισιόν κάνει καλά τη δουλειά της, παρότι δεν με ενδιαφέρει να την υποστηρίξω, αλλά πραγματικά πρέπει να πούμε ότι συνήθως κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήσταν πράγματι ε, σύντομη, κύριε Τόμψον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ε, για αυτά που είπατε, για την κοινοτομία ιδίως ήταν πολύ σημαντική η έκθεση που εξετάζει, που μελετά τη βιομηχανική δομή της Ευρώπης, γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται. Γιατί νομίζω και ο τίτλος αυτής της ακροάσης είναι λίγο παραπλανητικός. Δεν συζητάμε τώρα τη βιομηχανική πολιτική. Συζητάμε την πολιτική παραγωγής, την, την ε, ε, πολιτική βιομηχανικής παραγωγής Θέλω να είμαι λίγο προκλητική και να πω ότι μάλλον σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Στη, δεκαετία του 80 οι μετανάστες στο, Ευρω... στο Ενωμένο Βασίλειο ε, έκλεισαν, ε, ε μάλλον τα, τα ανθρακοριχεία και το Ηνωμένο Βασίλειο στράφηκε σε άλλο τομέα. Και όταν άκουσαν οι νέοι άνεργοι ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούν ε, από τη νέα, κυβέρνηση των νέων εργατικών, αυτοί δεν ευχαριστήθηκαν γιατί έπρεπε <laughs> από, γιατί έπρεπε να αφήσω αυτό που έκαναν. Τι έκαναν, έπαιζαν μουσική τι είναι πιο σημαντικό, η βιομηχανία pop music στην Αγγλία ή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Τι σημαίνει λοιπόν βιομηχανική παραγωγή. Μιλάμε μόνο για βιομηχανική πολιτική, ε, γιατί τότε πρέπει να μιλάμε και για την pop music. Γιατί ε, εγώ είμαι Δανία, πάνω από το 10, κάτω από το 10% των εργαζομένων ε, στη Δανία ασχολούνται με τη βιομηχανία, αλλά αυτή τη στιγμή ε, αυτή έχει μετακινηθεί στην Κίνα και αλλού. Και μιλάμε για ε, πρώτε ύλε. Δεν έχουμε πολλέ πρώτε ύλε. Η Αφρική έχει πολλέ πρώτε ύλε, αλλά στην Ευρώπη ζούμε καλύτερα, πιστεύω. Τι σημαίνει πρώτε ύλε, δεξιότητε. Και νομίζω είναι το, το καλό εργατικό δυναμικό. Αυτή η βιομηχανική παραγωγή που έχουμε μετακινήσει εκτός Ευρώπης, πιστεύετε ότι πρέπει να επιστρέψει. Πρέπει να αρχίσουμε πάλι να κατασκευάζουμε την Ευρώπη ή να πούμε πάει αυτό τελείωσε, ας πούμε η κλωστοϊφαντουργία. Εμείς σχεδιάζουμε, πολλούμε, κάνουμε το μάρκετινγκ, αλλά η παραγωγή γίνεται κάπου αλλού. Στην Κάνα, αν δεν κάνω λάθος πλέον. Αυτό μήπως πρέπει να το κάνουμε. Και νομίζω ότι αντιπροσωπεύεται κλάδους όπου υπάρχει ε, πολύ ανδρική απασχόληση. Πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε χώρο για τις γυναίκες εκεί, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Στο μέλλον να δούμε ότι το 75% του εργατικού δυναμικού ε, το 2020 στην Ευρώπη θα είναι γυναίκες. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Président.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 Uh, Το που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η χημική βιομηχανία δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, ε, δεν φοβάται τους ελέγχους, δεν φοβάται την ιχνηλασιμότητα. Ε, όμως είναι γεγονός ότι εμείς ε, εξαρτώμαστε πολύ από εισαγωγές αλλά και από τις εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο και επομένως ε, οι περιορισμοί στα σύνορα μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Βεβαίως εμείς δεν προτιθέμεθα καθόλου να μειώσουμε την ανάπτυξη οποιοδήποτε, οποιοδήποτε χώρας του κόσμου. Βεβαίω, οι νομοθετικέ ρυθμίσει, τα νομοθετικά πλαίσια είναι απαραίτητα, αλλά η χημική βιομηχανία αυτή τη στιγμή βλέπει πολλού νόμου να ξεπερνούν σύνορα Α πούμε μια μεγάλη ε, ε, βιομηχανία θα τα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα γιατί έχει και πόρου, έχει και τεχνογνωσία και έχει τη δυνατότητα να πάει και αλλού στον κόσμο. 96% τη χημική βιομηχανία όμως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να μαζέψουν τα πράγματά τους και ε, το εργοστάσιό τους και να φύγουν να πάνε αλλού. Ε, εξαρτώνται πολύ από αυτό το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και συγκρίνουν ε, διαρκώς ε, το τι κάνει η Ευρώπη με την ε, Βραζιλία, με την Ευρώπη, με την Ινδία, τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνουμε εμείς. I, I, I want to ask... Και εγώ σας ρωτώ. Εάν δούμε ότι η ενέργεια είναι πιο ακριβή στην Ευρώπη από ό,τι στις άλλες χώρες του κόσμου, εάν δούμε ε, ότι η βιομηχανία αυτόνομα και μεμονωμένα ε, εισάγει νέα μέτρα, τότε ε, θα είναι κανείς ανόητος εάν δεν προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Εάν ήδη πληρώνει κάποιος περισσότερα για τις πρώτες ύλες από κάποια άλλα μέρη του του δεν θα προσπαθήσει να αντιστρέψει την κατάσταση αυτή. Το θέμα της ενιαίας αγοράς ε, ετέθη. Ναι, η ενιαία αγορά είναι όντως ένα σημαντικότατο στοιχείο για τις ε, μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Βλέπω στο ανακοινοθέν στην ανακοίνωση, μάλλον ανέβλεπα στην ανακοίνωση Επιτροπής το θέμα της παγκοσμιοποίησης, της παγκόσμιας δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ θα έλεγα ας δώσουμε πρώτα τη δυνατότητα ευρωπαϊκής δράσης και ε, μετά να πάμε στην Ινδία ή στην Κίνα. Αναφερθήκατε, ε, κυρία μου, στην, ε, στο θέμα της καινοτομίας. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με ορισμένους τομείς περισσότερο από ό,τι με άλλους. Ε, ε, βεβαίως ε, η Επιτροπή λέει θέλω κάτι σχετικά με το νερό, τότε θα μιλήσω στην, ε, με τους υπεύθυνους βιομηχανίας του νερού. αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που σχετίζονται με το νερό. Υπάρχουν υδατοκαλλιέργειες, υπάρχουν και πρέπει να σας πω ότι η χημική βιομηχανία το προηγούμενο χρόνο έκανε μία ένα κοινό εγχείρημα ε, με τις εταιρείε που ασχολούνται με το νερό έτσι ώστε να δημιουργηθούν κάποιες ε, ε, συνέργειες για να βρεθούν λύσεις και για το πόσιμο νερό και για τις βιομηχανικές χρήσεις του νερού. Μέσω των συνεργειών λοιπόν μπορούμε να βελτιωθούμε. Εμείς δεν θέλουμε χρήματα, εμείς θέλουμε ένα καλό ανταγωνιστικό πλαίσιο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στον κόσμο. Και νομίζω ότι εδώ, από εδώ και στην ερώτηση της κυρίας Γκροστέτ, υπάρχουν αρκετά χρήματα για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για την καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε λίγα από τα ζητήματα που τέθηκαν και να μην σας καθυστερήσω. Ένα όμως από τα ερωτήματα ήταν ότι ε, αν η ευρωπαϊκή πολιτική πιστεύουμε ότι θα μπορεί να είναι καλή χωρίς ε, να ασχοληθούμε σοβαρά με την ε, απασχόληση. Είπα νομίζω ξεκάθαρα ότι πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και το, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ποια θα είναι η καλύτερη τοποθέτηση των επενδύσεων και συμφωνώ με αυτά που άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Τόμψον η επένδυση στους Ευρωπαίους εργαζόμενους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και η εξασφάλιση ότι πολλοί εργαζόμενοι θα έχουν ε, στη δουλειά ε, πρόσβαση στην ε, κατάρτιση και στην επανακατάρτιση θα αποτελεί σοβαρό βήμα προόδου στην ανάπτυξη της κοινοτομία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και στην ανάπτυξη νέων τομέων, νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Αναφέρθηκα στο θέμα του ε, φόρου των συναλλαγών. Όμως ε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνδικάτων αναπτύξαμε το θέμα. Ε, έχουμε μία έκθεση που πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσω νέο, της ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών μέσων. Επίσης, θέλω να συμφωνήσω με την ιδέα ότι δεν πρέπει να έχουμε ε, κλάδους που να χάνουν και να μολύνουν το περιβάλλον. Όλοι οι κλάδοι μπορούν να καινοτομήσουν και να εμπλακούν στο θέμα της καινοτομία και αυτό έχει σχέση και με την εφοδιαστική αλυσίδα. Και όσον αφορά την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης και την επιστροφή των βιομηχανιών, πρέπει να είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για τις παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς της Ευρώπης, έχουμε και στην Ευρώπη ειδικού τομείς όπου εκεί που δεν το περιμένει κανένας και η, η είναι ένας από αυτούς. Υπάρχει υπεροχή σε αυτό το τομέα, αριστεία όσον αφορά τα υλικά της κλωστοφαντουργίας και την ε, βελτίωση της απόδοσης της ενέργειας στη μεταφορά και, τον, μηχανημάτων. Δεν πρέπει λοιπόν να κοιτάμε ε, τους παραδοσιακούς κλάδους, αλλά να ψάχνουμε τους τομείς όπου μπορεί να υπάρξει καινοτομία. Και στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής ε, απασχόλησης, σαφώς τα θέματα του φύλου, της ισότητας των φύλων είναι σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το θέμα για τις ευρεσιτεχνίες. Πράγματι υπάρχει Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, αλλά βέβαια υπάρχουν και στις υπόλοιπε ε, χώρες οι ανάλογες υπηρεσίες, οπότε πρέπει να υπάρξει και μετάφραση και δήλωση στις αντίστοιχες υπηρεσίες, οπότε αυτό είναι δύσκολο ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά ακούστηκε το ερώτημα ποιους τομείς ε, πρέπει να προωθήσουμε για να επαναφέρουμε εδώ πέρα τις βιομηχανίες παραγωγής. Βεβαίως όχι εκεί πέρα όπου είναι φτηνή η εργασία και χρησιμοποιούνται πάρα πολλές πρώτες αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς που είναι ένταση εργασίας Δηλαδή έχουμε 150 με 200 εκατομμύρια κτίρια, κατοικίες στην Ευρώπη που θα πρέπει να ανακιστούν. Εάν δηλαδή γίνουν εδώ πέρα πολύ αυστηρέ οι προδιαγραφές για την θερμομόνωση, τότε θα έχει αυτό σημαντική επίδραση στην δημιουργία θέσεων εργασίας και το, τη μείωση του κόστου εργασίας. Οπότε ο τομέα επίσης ο άλλος είναι στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Επίσης αναφέρθηκε το τι γίνεται με τι διατάξει ε, για το διοξείδιο του άνθρακα, ποιοι είναι οι στόχοι του οποίου θέλουμε και εδώ πέρα πρέπει να το πω ξεκάθαρα από πλευράς προστασία του κλίματο Καλό θα ήταν να έχουμε πολύ δυνατούς ε, στόχους, υψηλούς στόχους, ε, στις οποίες, τις οποίες θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπε περιοχές του κόσμου. Από πλευράς βεβαίως ε, βιομηχανικής πολιτικής μπορώ να πω έτσι κάπως ηρωνικά πως όσο τόσο το καλύτερο να έχουν χειρότερο στόχους οι άλλες περιοχές γιατί έτσι θα έχει προβάδισμα η Ευρώπη γιατί σημαίνει πως θα ε, είναι χαμηλότερο το ενεργειακό κόστος και θα γίνει η Ευρώπη ανεξάρτητη από τις εισαγωγέ ενέργειας, ε, από εισαγωγές πρωτονολών όπως το Νεοδήμιο και τα λοιπά και ταυτόχρονα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογική της ικανότητα για να προωθήσει προς τον Οπότε αυτή είναι η σύστασή μας για το τι θα πρέπει να προωθήσουμε και να έχουμε βεβαίως φιλόδοξους στόχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Μανολίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος. Θα ήθελα εγώ να επανέλθω στην αρχική μου τοποθέτηση για την ε, εμπειρία ορισμένων κοινωνιών και κάποιους κινδύνους γιατί αναφέρεται πάρα πολύ ο κίνδυνος στην Ευρώπη ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ότι στο παρελθόν όπου λίγοι μόνο μπορούσαν να εκφράσουν την άποψή τους αλλά βεβαίως να επανέλθουμε στα ερωτήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά Μιλάμε για τις ε, πολιτικές ε, προοπτικές. Οπότε όσοι θέλουν να χαράξουν στρατηγική πρέπει να δουν ε, και το τι θα κάνουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε παραγωγή στην Ευρώπη και μία πρόταση είναι βεβαίως να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση και να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα λεφτά γιατί σπαταλούνται τόσα πολλά στην Ευρώπη μέσω κακής ε, διοίκησης και διαχείρισης και βεβαίως να έχουμε και εταιρικέ σχέσεις όχι μόνο δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αλλά και άλλες για να μπορέσουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Η πραγματικότητα βεβαίως ε, είναι πάντα κάπως διαφορετική Ίσως υπάρχει το μοντέλο της κοινωνικής ε, Ευρώπης ε, σε αντίθεση με τη ΣΥΠΑ και του τι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν σημαίνει βεβαίως πως το ένα σύστημα μπορεί να μεταφερθεί αυτούσιο στο άλλο. Και βέβαια το θέμα είναι αν θα ήταν επιτυχημένο ένα αμερικάνικο μοντέλο εδώ πέρα. Ενώ άλλοι λένε πως ε, τα συνδικάτα είναι ανταγωνιστικά με τους ε, εργοδότες. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είχα πει στην αρχή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν την ε, Ευρώπη. Να σας αναφέρω και τα αυτοκίνητα, τα, τα Dacia, που είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία που φτιάχνει τα αυτοκίνητά της στην Ευρώπη. Είναι Συχά στον κύριο Ενέν, το ζήτημα έχει λυθεί. Μιλάμε τώρα για μια εταιρεία με τριπλάσια ή με τριπλάσιο ήδη δυναμικό. Σημασία έχει λοιπόν να παράγουμε στην Ευρώπη ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα βρίσκεται η παραγωγή. Η παραγωγή είναι η λύση στην Ευρώπη. Μιλάω και για τις δημιουργικέ βιομηχανίε και εκεί πέρα έχει να πει κάτι και η Ευρώπη. Οπότε, τελειώντα. θα ήθελα να πω πως ε, εάν συνεργαζόμαστε πιο αρμονικά νομίζω θα έχουμε καλύτερη παραγωγική δομή στην Ευρώπη και θα αποφύγουμε πάρα πολλές παγίδες και προβλήματα. Αλλιώς θα έχουμε χειρότερα προβλήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Του συναδέλφου εδώ πέρα στο Προεδρείο. Νομίζω πως είχαμε συνένεση, θέλουμε όλοι μαζί να κινηθούμε και βεβαίως και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με όλα αυτά να κινητοποιηθούν για να έχουμε καλύτερη δημιουργία πλούτου στην Ευρώπη και να έχουμε και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος σε κάποια σημεία στην ανακοίνωση της Κομισιόν ε, στο ζήτημα της συμπερίληψης ε, των κοινωνικών εταίρων. Είμαι επίσης πεπισμένος και αυτό το είπε και η κυρία Γκροστέτ, ε, η βιομηχανική πολιτική δεν θα πρέπει να είναι μόνο βιομηχανική πολιτική, αλλά ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, κατά το οποίο θα φαίνεται και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο των κρατών μελών, ότι δηλαδή όλοι μαζί έχουμε ένα κοινό στόχο και ο στόχος αυτός ε, είναι αηφόρος ε, ε, ανανέωση της βιομηχανικής μας βάσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και θα έχουμε την έκθεση βεβαίως στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε. Θα περάσουμε στα επόμενα βήματα. Κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μας που μας δίνεται η δυνατότητα να υποδεχτούμε την Επίτροπο για την κλιματική αλλαγή, την Κόνι Χέντεγκάρτ. Κύριε Επίτροπε, σας είμαστε ιδιαίτερως ευγνώμονες που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ήρθατε σε μια περίοδο που προετοιμαζόμαστε για την διάσκεψη της Κανκούν για την κλιματική αλλαγή. Είμαστε μια επιτροπή η οποία έχει εμπλακεί σημαντικά στην ε, προετοιμασία αυτή. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή σας για μας και σας δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους μπορέσαμε να βρούμε ένα κατάλληλο χρόνο για να έρθω εγώ σε εσά. Θα πω δύο λόγια για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις όπως μου ζήτησε η, ο πρόεδρος, αλλά θα μπορέσουμε ελπίζω να συζητήσουμε τα άλλα θέματα της αρμοδιότητάς μου. Θα πω όμως δύο λόγια πρώτα για την κατάσταση ε, των διεθνών διαπραγματεύσεων. Αυτό το Σάββατο ε, επέστρεψα από το pre-COP στο Μεξικό. Είναι η τελευταία ε, ευκαιρία να κάνουμε μια διαπραγμάτευση πριν την διάσκεψη αυτή καθεαυτή, η οποία ε, διάσκεψη θα αρχίσει αυτό το μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 10 Δεκέμβρη. Τι περιμένουμε από αυτή τη διάσκεψη. Όταν το Μάρτιο η Κομισιόν πρότεινε ότι δεδομένου ότι τίποτα το καινούριο δεν είχε προκύψει ούτε από το Πεκίνο, ούτε από πολλές άλλες πρωτεύουσες μέχρι την Κοπενχάγη την Άνοιξη, πρέπει να επιδιώξουμε μία προσέγγιση βήμα με βήμα, προς βήμα. Φαίνεται ότι όλοι πλέον συμφωνούν με αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε μέχρι την Κανκούν να καταλήξουμε στην νομικά δεσμευτική συμφωνία, όχι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξέρετε ήδη από την Κοπενχάγη είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε, ακόμα είμαστε έτοιμοι, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέρασε την νομοθεσία από τη Γερουσία, δεν μπορούμε λοιπόν, δεν είχαμε δυνατότητες από το Πεκίνο κλπ. κλπ. Άρα μοιάζει ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη ότι πλέον στην Κανκούν πρέπει να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε ένα ουσιαστικό πακέτο. Τι σημαίνει αυτό. Να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε για ένα πλαίσιο που αφορά τα δάση. Να σταματήσουμε την ε, αποψήλωση των δασών. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα στην Κοπενχάγη. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την προσαρμογή, ένα πλαίσιο προσαρμογής. Και επίσης ένα πλαίσιο τεχνολογίας σχέση με τον οποίο φαίνεται ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάσταση απόψε. Φυσικά, οι ανεπτυγμένε χώρες εννοείται ότι πρέπει να ε, δεσμευτούν, μάλλον να ε, εκπληρώσουν τις οικονομικές τους δεσμεύσεις. Και τώρα, από, οικονομική σκοπιά, από ευρωπαϊκή σκοπιά, θέλουμε και εμείς να γίνει πρόοδο στον τομέα του MRV. Ακούγεται τεχνικό και είναι. Δηλαδή, το θέμα είναι πώς θα αναθέσουμε και θα επαληθεύσουμε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Είναι όμως σημαντικό για τη διαδικασία. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεσμευτούμε κάτι, ε, για κάτι, αλλά να μην μπορούμε να το επαληθεύσουμε. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για μια διαφάνεια που θα πρέπει να εξασφαλιστεί στη διαδικασία αυτή όλες, δεν είναι όλοι εξίσου ενθουσιώδεις για τη διαφάνεια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο τομέας αυτός είναι δύσκολος, όμως εκεί προχωρούμε. Κάναμε πρόοδο στη Συμφωνία της Κοπερχάγης και άρα πρέπει με την Κανκούν να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Και το τελευταίο που θέλω να πω αφορά τις αγορές του άνθρακα από σκοπιά ευρωπαϊκή αλλά και από παγκόσμια σκοπιά πρέπει να καταλάβουμε γιατί πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα των CTM. Δεν, μπορούμε, δεν πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό, αλλά είναι ένα θέμα για την Κανκούν. Στην Κανκούν πρέπει να πετύχουμε ένα ισορροπημένο πακέτο. Δηλαδή δεν θα κάνουμε μόνο τα εύκολα και όλα τα δύσκολα να τα αφήσουμε για άλλη φορά πρέπει να είναι, υπάρχει ισορροπία και αυτό γι' αυτό πιέζουμε εμείς τις διαπραγματεύσεις. Τέλος, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις πρέπει να πω ότι γίνεται και αυτή η συζήτηση. Αν η ε, Ευρώπη θα ε, αναλάβει μια δεύτερη δέσμευση σε σχέση με τον πρωτόκολλο του Κιώτο. Πέρυσι κατηγορήθηκε ότι θέλουμε να εξαφανίσουμε το Κιώτο. Πάντα το θεωρούσα περίεργο, διότι όλες οι εσωτερικές πολιτικές Ευρώπης στηρίζονται στις αρχές του Κιώτο. Γιατί λοιπόν να μας ενδιαφέρει να το εξαφανίσουμε, να το σκοτώσουμε. Λέμε λοιπόν τώρα, όχι, είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, υπό όρους όμως. Διότι θα πρέπει και οι άλλοι να δεσμευτούν. Αυτός είναι ο ένας όρος. Και Κάποιες από τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος του Κιώτο είναι αρκετά μπερδεμένα και τεχνικά, θα επανέλθουμε. Υπάρχουν όμως κάποιες αδυναμίες που δεν εξασφαλίζουν την ε, περιβαλλοντολογική ακαιρεότητα, πρέπει να πάνε εξεταστούν. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς δεσμευτήκαμε εν ώψη του Κιώτο, κάναμε αυτά τα οποία ε, υποσχεθήκαμε, κάναμε και παραπάνω, έχουμε ε, λοιπόν πρόβλημα, θέλουμε και οι άλλοι να κάνουν αυτά που υποσχέθηκαν. Αυτό ζητάμε, αυτό θεωρούμε σημαντικό, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και τότε θα σας πει, όταν επιστρέψετε από το, ήρθατε από το Μεξικό, όταν επιστρέψετε το Μεξικό, κυρία Επίτροπε, και έχουν όλα ξε, ε, ξεχαστεί. Κοιτάξτε, προκαταρτικά υπήρχε καλή θέληση, επικοδομητική διάθεση, τα έχω δει όλα αυτά σε τέτοιες περιστάσεις και είναι καλά. Αλλά στην ουσία είναι η ουσία βρίσκεται στο αν και κατά πόσον όταν φτάσουν όλοι στην Κανκούν θα κάνουν τους απαραίτητους συμβιβασμούς. Αυτό θέλουμε να επιτευχθεί, θέλουμε να προωθήσουμε τα πράγματα και σας διαβεβαιώνω. Φροντίζουμε να καταλάβει η Ευρώπη πόσο σημαντικό είναι να μιλάει με μια φωνή. Το μήνυμα της Ευρώπης και των κρατών μελών πρέπει να είναι το ίδιο αν θέλουμε να μας ακούσουν και αν θέλουμε να έχουμε επιρροή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα αφήσω τώρα την Κανκούν και το τι θα γίνει εκεί και θα επανέλθουμε σε διάρκεια της συζήτησης. Θα ήθελα τώρα, ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια άλλα ζητήματα της αρμοδιότητός μου, τα οποία νομίζω ενδιαφέρουν και την Επιτροπή σας. Υπάρχουν κάποιες δράσεις σχετικές με το κλίμα στο πρόγραμμα εργασίας του 2011 της Επιτροπής που υιοθετήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Βασική προτεραιότητα είναι η εφαρμογή της Ατζέντα για το 2020 και των βασικών πρωτοβουλειών, μεταξύ των οποίων και η πρωτοβουλία για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Για να το επιτύχουμε αυτό και το μέλλον με χαμηλό άνθρακα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν όλες αυτές τις πολιτικές, δηλαδή ενέργειες κλιματικής αλλαγής μεταφορών και περιβάλλοντος, οριζόντιες, να μην κοιτάω καθένας το χαρτοφυλάκιό του, αλλά η Κομισιόν συνολικά να βλέπει τα πράγματα πιο οριζόντια. Το πρόγραμμα εργασίας Κομισιόν για το 2011, άρα προβλέπει μια συνολική προσέγγιση που ορίζει το πώς η ενέργεια, οι μεταφορές και η οικονομία χαμηλού άνθρακα θα μετασχηματίσουν και θα μεταμορφώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία μέχρι το 2050. Αυτό θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο ένα οδικό χάρτη μέχρι το 2050 που ετοιμάζουν οι υπηρεσίε μου, αλλά και τη λευκή βίβλο για τις μεταφορές και τον ενεργειακό χάρτη για το 2050, το οποίο θα παρουσιάσουν οι Επιτροπή Έτσιγκερ και Κάλλας. Όλα αυτά δεν θα ενισχύσουν μόνο την οικονομία μας, ήδη προσφέρουν ευκαιρίες σήμερα. Οι θέσεις εργασίας ε, αυξάνονται κατά 7% το έτος από το 2000 και εδώ και έχουμε μια πραγματική προοπτική εκατομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020 θα μπορέσουμε έτσι να πάμε πέρα από το στόχο μείωσης κατά 20% και την προετοιμασία μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα. Σύμφωνα με τις διεθνείς μας δεσμεύσεις ότι θα οδηγηθούμε σε μείωση 95% μέχρι το 2050 σύμφωνα και με το στόχο των δύο βαθμών. Στοχεύουμε την άνοιξη του 2011 να υιοθετηθεί και να δημοσιευτεί αυτό ο χάρτης και θα έχουμε και τα ενδιάμεσα βήματα για να φτάσουμε εκεί, κάτι το οποίο υπονοεί πως θα συμπεριλάβουμε στόχο για το 2030. Θα ξέρετε πως από την πλευρά του επενδυτή το 2020 είναι αύριο, οπότε οι επενδυτές στον τομέα τη ενέργεια σκέφτονται πέρα από το 2020, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα για το ποιοι θα είναι οι στόχοι μας για το 2030. Νομίζω πως αυτό θα επηρεάσει και την συζήτηση για τους βραχυπρόθεσμους στόχους, γιατί αν ξέρουμε ποιος είναι στόχος για 2030 και 2050, μπορούμε να δούμε πως εάν χαλαρώσουμε μέχρι το 2020, κινδυνεύουμε να είναι δύσκολα τα πράγματα για μετά το 2020. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουμε την ανακοίνωσή μας, αυτή που βγάλαμε το Μάιο, για το κόστος και το όφελος και τις προκλήσεις του να πάμε πέρα από το 20%. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να αναλύσουμε ε, σε επίπεδο κράτους μέλους ε, αυτά τα οποία έχουμε σε ευρωπαϊκό στόχο. Θα πω επίσης πως η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τι θα προκύψει από πλευράς Κοινοβουλίου Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό εκεί πέρα και ενδιαφέρον είναι να δούμε το εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στο κοινοτικό προϋπολογισμό για να στοχεύσουμε με τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Υπάρχουν πολύ εύκολοι στόχοι στα κράτη-μέλη όταν μιλάμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά ειδικά για τα νέα κράτη-μέλη πιθανότερο θα είναι να επιτύχουμε αυτούς τους εύκολους στόχους αν έχουμε κάποια βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Τέλος, να πω λίγα πράγματα για κάτι άλλο. Η συγκριτική αξιολόγηση, ξέρω πως ενδιαφέρει την Επιτροπή σας, όπως ξέρετε, είχαμε, κάνει, είχαμε ξεκινήσει ένα σχετικό εγχείρημα για τους τομείς οι οποίοι κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τη διαρροή άνθρακα για να χαθούν θέσεις εργασία σε άλλα μέρη του κόσμου. 52 κλάδοι θα εξαιρεθούν και ε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό το εγχείρημα. Ξέρω πως θα σας προσεγγίσει η βιομηχανία. Νομίζω πως πολλοί κλάδοι αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιημένοι αυτή τη στιγμή. Η βιομηχανία αναγνωρίζει πως είναι δύσκολο αυτό. ήταν η Κομισιόν που είπε πως έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα. Πέρσι η Κομισιόν πρότεινε να κάνουμε πληστηριασμό. Αλλά το Κοινοβούλιο, ε, συγγνώμη τα κράτη-μέλη και η βιομηχανία προτίμησαν αυτή την αξιολόγηση και ορίσαμε κάποια κριτήρια για το πώς θα γίνει. Τώρα ε, δεν ήταν εύκολο αυτό, ήταν μια περίπλοκη διαδικασία και ελπίζω να αντιλαμβάνεστε πως ε, πρέπει να είμαστε συνεπείς στην αξιολόγηση αυτή. Δεν γίνεται με τον ένα τρόπο για τον ένα κλάδο και με άλλο τρόπο για άλλο κλάδο. Πρέπει τουλάχιστον να είμαστε συνεπείς με την οδηγία. Νομίζω πως τώρα οι περισσότεροι κλάδοι θεωρούν πως είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Ανέβαλα τη δημόσια διαβούλευση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές για πολλούς μήνες για να λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες της βιομηχανίας, αλλά πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τις αρχές. Γνωρίζω πως αυτό θα σας ενδιαφέρει. Θέλω να τελειώσω λέγοντας πως είναι κρίσιμο να αποδεχτούμε πως θα είναι τεχνική παραπολιτική αυτή η υπόθεση και ό,τι πάρουμε από τον ένα κλάδο ή δώσουμε σε ένα κλάδο θα πρέπει να αφαιρεθεί από αλλού. Γι' αυτό συμβουλή μου είναι να μην γίνει πολιτικό το ζήτημα, γιατί υπάρχουν αυστηρά κριτήρια στην οδηγία και αν δεν τα τηρήσουμε θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα μπω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες, νομίζω πως κυκλοφορεί από πλευράς βιομηχανίας ε, ε, ξέρετε πως τα πράγματα έχουν ένα ιστορικό. Αυτά νομίζω καλό είναι να δεχτώ ερωτήσεις, ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για την συνοπτική αναφορά σας στις διπλωματικές προσπάθειες στα πλαίσια της ε, Κανκούν και για την στρατηγική σας για τον επόμενο χρόνο και πέραν. Πολύ ενδιαφέρουσα για μας ε, η παρουσίασή σας αυτή. Και σημαντική ε, συμβολή στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Επίτροπε. Για να υπάρξει ένας προγραμματισμός που θα συμπεριλαμβάνει και μια αναπτυξιακή πολιτική μέχρι το 2020. Κάτι το οποίο βέβαια υπήρχε στην αρχική μας ε, πρόταση για την αηφόρο ενέργεια, καθώς στόχος μας ήταν η Κομισιόν να υποβάλει αυτό το σχέδιο αϊφορουμίωσης του 2007 ήταν τότε ένα σοκ αυτό ε, για τους Ευρωπαίους ε, λομπίστες οπότε θα πρέπει μέχρι το 2020 να έχουμε 20% ε, ανανεώσιμη ενέργεια αλλά θα πρέπει να πάμε και πέρα από αυτό πότε Η λογική συνέπεια του δεσμευτικού αυτού 20% είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα έχουμε πλειοψηφία, αλλά η Κίνα έχει ένα στόχο 20% μέχρι το 2011 και άλλο 17% ε, βεβαίως μιλάμε για ε, ένταση ενέργειας. Οπότε όταν μιλάμε για ανάπτυξη, νέες μεθόδους ε, κτλ. θα πρέπει να μείνουμε τουλάχιστον στο επίπεδο της Κίνας. Αλλά αν δεν μπορούμε να έχουμε δεσμευτικούς στόχους θα μπορέσουμε να παραμείνουμε στο επίπεδο της Κίνας. Μπορούμε να είμαστε first mover, τι Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ μονάχα τρία λεπτά ανασυνάδελφο για τις ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε κυρία Επιτροπέ. Δύο ερωτήσεις. Μία για το AAUs εάν δώσουμε, αν δώσαμε κάποια εκατομμύρια ε, στην Πολωνία και σε άλλες χώρες ε, το 2008, με εκπλήσει που οι ίδιες χώρες επανέρχονται τώρα και κατά κάποιο τρόπο ε, δυναμητίζουν την Συμφωνία του Δεκεμβρίου 2008. Εάν θέλουμε όμως να διατηρήσουμε τις συμφωνίες Κιώτο Μπορείτε να μου, πείτε πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό από τεχνικής απόψεως. Και τι θα είχαμε, μια εξοικονόμηση 60-70-80 εάν μείνουν στο σύστημα. Δεύτερον, στην Επιτροπή μας εδώ ακούμε ένα σωρό επιχειρήματα από πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κερδίζουν πολλά χρήματα. και που δεν συμφωνούν με το 30%. Στη Γενική Διεύθυνση Κλίματος έχετε αναλύσει τις ε, βιομηχανίες ε, οι οποίες θα μπορούσαν να κερδίσουν την αλλαγή του κλίματος. Πώς μπορείτε λοιπόν να ε, ορίσετε την ανταγωνιστικότητα, γιατί βρίσκω στην Επιτροπή μας μερικές φορές εδώ δίνουμε πολύ συσταλτική εμπειρία και έχουμε βεβαίως ένα 6-7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που είναι συνδεδεμένο με την ένταση ενέργειας και ενδεχομένως εμείς ε, βλέπουμε μόνο ε, κάποια δέντρα και χάνουμε τη γενικότερη εικόνα που αφορά τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και βεβαίως πολλοί ακόμα και οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να κερδίσουν από αυτήν την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συνεχίζοντας τα λεγόμενα του συναδέλφου Τούρμες, ε, οι αξιολογήσεις, οι εκθέσεις ε, υπάρχουν για να καταδείξουν ότι η φιλοδοξία, η τη φιλοδοξία όσον αφορά το περιβάλλον και την, το, τις αλλαγές, κλιματικές αλλαγές, χρήση ανανεώσεων πηγών ενέργειας μπορεί να κοστίσει ακριβά στην κοινωνική Ευρώπη. Πώς μπορούμε να περάσουμε λοιπόν το σωστό μήνυμα στην Ευρώπη, στις ε, χώρες, έτσι ώστε να πείσουμε τους, ε, τις χώρες μέλη γιατί ακόμα και εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε μάλλον την τάση να οπισθοδρομούμε ε, και να ζητάμε τελικά λιγότερο όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, όσον αφορά το περιβάλλον. Τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να πείσουμε τους συναδέλφους στις χώρες μας ότι ότι οι μελέτες που υπάρχουν μπορεί να έχουν ένα καλό οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα. Δεύτερο ζήτημα. Τι γίνεται με την διαφάνεια της χρηματοδότησης των κρατών μελών όσον αφορά την πρώιμη χρηματοδότηση στην ε, Συμφωνία της ε, Κοπενχάγης και στη διαπραγματεύση της Κανκούν. Τελικά δηλαδή γίνεται σεβαστή η αρχική συμφωνία, δηλαδή ε, κρατική βοήθεια προσθετική και είδη χορηγίας και επίσης ποια είναι η συνέχεια που προτίθεστε να δώσετε στην πολύ καλή ανακοίνωση που είχατε κάνει πριν από μερικούς μήνες και που έλεγε ε, πως ε, πραγματικά η Ευρώπη θα κερδίσει αν περάσει το 30%. Κύριε Σοντή, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ορίσατε κυρία Επίτροπε. Έχουμε την αίσθηση σήμερα ότι ο διάλογος σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται δύσκολος και όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και όσον αφορά το περιβάλλον. Αν θέλουμε να είμαστε ορθολογιστές ε, ε, και αν θέλουμε να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο της, ε, του Κιώτο που βεβαίως δεν είναι δεσμευτικό απέναντι στις ΗΠΑ που δεν το έχουν υπογράψει και πέρα από την χρήση εργαλείων που υπάρχουν, μήπως αναπεριοχές του κόσμου, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νότια Αμερική. Ε, δεν θα έπρεπε, λέω, να απομονώσουμε τις υπήρους που δεν θέλουν να μας ακολουθήσουν σε αυτό το βηματισμό και στους ε, χώρους στους οποίους ε, οι πολίτες αποφάσισαν και οι χώρες αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτές τις αρχές. Δεν θα έπρεπε να απομονώσουμε τις άλλες χώρες έτσι ώστε τουλάχιστον στις ε, χώρες μας να έχουμε ενισχυμένες ε, ε, συμφωνίες πολυμερείς ή διμερείς συνεργασίες, ας πούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, Νότια Αμερική, με κάποια ενδεχομένως νομοθετικά εργαλεία αλλά κυρίως να είμαστε βέβαιοι ότι ε, και οι κοινωνικές ρήτρες και οι περιβαλλοντικές ε, ρήτρες ε, θα καλύπτονται. Να, να δημιουργήσουμε δηλαδή με, κατά κάποιο τρόπο ζώνες ελεύθερων συναλλαγών με περιβαλλοντικό περιεχόμενο ακολουθώντας κάποιους ε, κάποιες καλές συνεργασίες και απομονώνοντας ε, περιοχές του κόσμου όπως ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα. Γιατί στην ουσία όλοι λέμε μπράβο τι ωραία που τα συζητάμε αλλά δεν υπάρχει τίποτα αναγκαστικό και υποχρεωτικό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χόλ. Um, Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτα απ' όλα, αναφέρατε πως η χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική για να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στην Κανκούν. Εγώ ανησυχώ, γιατί από όσο ξέρω, η πρώτη δόση των χρημάτων 2010-2012 δεν έχει πληρωθεί. 2,4 δισεκατομμύρια από τα 7,2 που έχει δεσμεύσει η Ένωση. Πότε θα τα δούμε αυτά τα λεφτά γιατί αυτό μπορεί να είναι ένα εμπόδιο ε, από πλευράς αναπτυσσομένων χωρών. Δεύτερον, τι διαβεβαιώσεις μπορούμε να δώσουμε στι αναπτυσσόμενε χώρες πως τα χρήματα αυτά θα προσθεθούν στην αναπτυξιακή βοήθεια. Γιατί οπωσδήποτε οι αφρικανικές χώρες παραπονιούνται πως τα λεφτά φύγανε από την υγεία Κατά ε, το οποίο βεβαίω δεν είναι ικανοποιητικό κατά την απόψή του. Δεύτερον, για τον, καθαρό, για τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης αναφέρατε το θέμα των στρεβλώσεων. Ξέρω πως υπάρχουν κάποια αέρια τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση πολλαπλάσια του διοξιδίου του άνθρακα και αυτό δημιουργεί κάποιες στρεβλώσεις και γενικότερα ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης πάει στην Κίνα και στην Ινδία, οι οποίες είναι χώρες που το χρειάζονται λιγότερο, είναι ήδη τεχνολογικά προοδευμένες και σπάνια πάει κάτι στην Αφρική. Νομίζω τώρα είχαμε μια αιωλική εγκατάσταση στο πράσινο ακροτήριο, αλλά είναι ένα από τα λίγα που πήγε στην Αφρική. Και τέλος, για να περάσουμε στο 30%, τι κινήσεις βλέπετε στο Συμβούλιο και σε ποιο βαθμό μπορούμε να περάσουμε το μήνυμα πως στο τωρινό πλαίσιο, στην τωρινή οικονομική κατάσταση μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο έτσι εύκολα. Ειδικά εάν τεθεί αυτός ο στόχος 20% ε, ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ. Αποδοτικότητας. Ευχαριστώ κύριε Καρβάγια. Thank you very much, Commission, for very detailed... Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την λεπτομερή περιγραφή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο ανέφερε και η συνάδελφος για τον μηχανισμό αυτών καθαρής ανάπτυξης. Γιατί αυτό είχε σχεδιαστεί και ως μέσο ανάπτυξης για έργα τα οποία θα μείωναν το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά θα είχαν και θετικές επιπτώσεις σε αυξόμενες χώρες. Ε, κατά βάση χρησιμοποιήθηκαν για βιομηχανικά αέρια. Καταστροφή δηλαδή εργοστασίων στην Ινδία και στην Κίνα και γύρω στο 8 και 9% των αδειών είναι από αυτά τα έργα. Δηλαδή είχαμε μεταφορά χρημάτων από την Κίνα και στην, στην Κίνα και στην Ινδία. Ε, δεν ήταν αυτός ο στόχος. Το ερώτημά μου είναι να επανασχεδιαστεί ο μηχανισμός αυτός. Αλλά ανησυχώ για το μέλλον. Υπάρχει ένας τρόπος να αποφευχθεί το ότι οι άδειε αυτές θα ε, συμπεριληφθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Υπάρχει κάποιο τρόπο. Γιατί κατά την άποψή μου συμπεριλήφθησαν κάποια έργα που δεν πλήρωσαν όλες τις ε, συνθήκες. γιατί δεν είχαν όλα τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε, δηλαδή να είναι θετικά για τις χώρες και να παρουσιάσουν ανάπτυξη κτλ. Βλέπετε λοιπόν κάποια διέξοδο έτσι ώστε η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να κάνουν κάτι με τις άδειε που προκύπτουν από αυτά τα έργα του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κυρία Ντελκαστήγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που ήρθατε σήμερα. εκ ε, μου προσωπικά αλλά και εκ μέρους της ομάδας μας σας ευχαριστώ θερμά. Πιστεύω ότι η συνάντηση της Κανκούν αποτελεί ευκαιρία για να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Αντίθετα με αυτά που συνέβησαν στην Κοπενχάγη, όπου είχαμε πολλές προσδοκίες. Τώρα είμαστε προσγειωμένοι. Και στην ουσία ψάχνουμε να βρούμε τις πραγματικές δυνατότητες επιτεύξης στόχων. Καλό πράγμα η φαντασία γιατί μας κινητοποιεί αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες που, αν μας επιτρέπουν να πετύχουμε ένα στόχο. Και υπάρχουν αυτοί οι στόχοι της Κανκούν που πιστεύω ότι εντάσσονται πολύ καλύτερα στην πραγματικότητα που επικρατεί σε αυτόν τον κόσμο πως ε, οι διάφορες χώρες, δηλαδή αυτές που κάνουν τις βασικές εκπομπές, ε, που είναι οι βασικοί ε, παράγοντες εκπομπών, θα ενταχθούν. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε σχέση με το πού πηγαίνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε η Επίτροπος ότι το 2020 είναι εδώ. Πράγματι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το 2030. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αρχίσουν να κάνουν ε, προγνώσεις, στρατηγικές, ε, αναπτυξιακές πορείες. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει από τώρα το 2030. Θεωρώ ότι το 30% είναι δυνατόν να εισαχθεί το ταχύτερο δυνατόν. Εγώ για να είμαι ειλικρινής πιστεύω ότι θα είναι σοβαρό σφάλμα αν ξεκινήσουμε ε, στο πλαίσιο αυτής της σοβαρής οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε, αντί να ε, ασχοληθούμε με την αποτελεσματικότητα των ε, αποφάσεων που έχουμε ήδη ληφθεί, να ασχολούμαστε με το να τηρηθούν οι στόχοι δηλαδή που έχουμε ήδη θέσει για να μην προσπαθούμε να επιτύχουμε υψηλότερους στόχους. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις να ε, κινηθούν σε ένα τόσο ευρύ ορίζοντα. Από οι τεχνολογικές προόδοι θα επηρεάσουν και τους στόχους που θέτουμε. Κάποια στιγμή ίσως μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα γρηγορότερα. γιατί η τεχνολογική ανάπτυξη προχωρεί. Σημασία λοιπόν έχει αυτό που θα αποφασιστεί στα ε, διεθνή θεσμικά όργανα και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κάτι το προσγειωμένο. Δεν θα πρέπει να προτρέχουμε και να ξεχνάμε την πραγματικότητα. Το σύστημα που έχουμε για την ε, αξιολόγηση αυτών που έχουμε για την επίτευξη των στόχων εκπομπών. Σημασία έχει να μας απασχολήσει σε συνεργασία με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα επιδιώκουν καλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη χρήση, τεχνολογίες που θα είναι αποτελεσματικές σε σχέση με την ε, κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κ. Καζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση προθέσεων αλλά έχω την εντύπωση πως στον τομέα της ε, κλιματικής αλλαγής απουσία ενός παγκοσμίου συστήματος πρέπει να έχουμε κατά νου οι προσπάθειες της Ευρώπης μόνο πάντα δεν θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Προφανώς, εάν η Ευρώπη είναι το 12% των εκπομπών, 20% αυτού είναι 3%. Οπότε ούτε και το 30% θα επιτύχει τους γενικότερους στόχους επιπλέον. Θεωρώ πως ε, πρέπει να δούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε διάφορους ε, τομείς. Ανέφερε η Επίτροπος στα δάση σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα μπορούσα να πω πως η χώρα μου φυτεύει δέντρα τα τελευταία 20 χρόνια. Η δασοκάλυψη έχει αυξηθεί κατά 3 με 4% ήδη. Νομίζω 30% δασοκάλυψη είναι χαρακτηριστική περίπτωση η Πολωνία για χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Οπότε η απορρόφηση του άνθρακα είναι σημαντική. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα δάση και το έδαφος, να δούμε το χούμους, το στρώμα αυτό του εδάφους. Καθώς <coughs> υπάρχει ήδη αντίκτυπος ε, από την ποιότητα των εδαφών, εάν αυξηθεί το ποσοστό του χούμου στο ε, έδαφος ε, συνεισφέρουμε στην απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα και αντιστρέφεται η τάση η οποία είναι να καταστρέφεται το έδαφος ε, το οποίο υπάρχει. Επίσης θέλω να ρωτήσω την κυρία Επίτροπο για το τι γίνεται με την επιτροπολογία και την συγκριτική αξιολόγηση, γιατί η βιομηχανία μας λέει πως Το φυσικό αέριο είναι το μόνο σημείο αναφοράς. Πολλοί μας λένε, ειδικά επενδυτές εκτός Ευρώπης, σκέφτονται το κόστος και σκέφτονται να πάνε την παραγωγή εκτός Ευρώπης. Τη στιγμή την οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 5,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Δεν μου φαίνεται και πολύ σωστό αυτό. Η International Paper είναι μία από τις εταιρείες οι οποίες κρούει τον κόμμα του κινδύνου. Και μετά κάτι για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τούρμες το 2008. Δεν είδαμε δισεκατομμύρια στην Πολωνία εμείς, αλλά επιτύχαμε πάρα πολλά ε, όσον αφορά το Και είχαμε και αναγνώριση για αυτές μας τις ενέργειες. Επίσης πρέπει να έχετε κατά νου το τι συνέβη στην προενταξιακή διαδικασία. Πολλές θέσεις εργασίας έφυγαν από την Πολωνία και μετατοπίστηκαν, αν θέλετε, στα υπάρχοντα κράτη-μέλη. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Πριν από 20 χρόνια ε, εμείς κάναμε ένα δημοψήφισμα για την πυρηνική ενέργεια και απορρίψαμε την πυρηνική ενέργεια στην Πολωνία. Αλλά αυτό το σκέφτομαι τώρα στο πλαίσιο του, του πυρηνικού τρένου. Δεν ξέρω, αν είχαμε μια, λάβει μια διαφορετική απόφαση, να μην είχαμε έλλειψη ενέργειας αυτή τη στιγμή. Είμαστε χώρα που έχει άνθρακα, αποθέματα άνθρακα, θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε και θέλουμε και να διατηρηθούν και οι θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και εγώ. Και ε, με συγχωρείτε που δεν είπα σωστά το όνομά σας. Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Λάγκεν. Äh, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την εικόνα τη γενική μας δώστε και για το ότι ήρθατε. Δεδομένων των πολιτικών εξελίσεων θαυμάζω την αισιοδοξία σας, είναι θετικό. Αλλά θεωρώ πως από την Κοπενχάγη και με βάση τα όσα συνέβησαν σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου δεν είχαμε καμία πρόοδο έχουμε συνθήκες οικονομικές οι οποίες επιδεινώθηκαν και μετά τις ε, εκλογές της ΕΠΑ όπου τώρα και η ήπια νομοθεσία των ΕΠΑ αποσύρεται από πλευράς Ομπάμα. Οπότε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Και να μην ξεχνάμε και τις ε, το νομισματικό πόλεμο είπα Κίνας, που θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις ε, στην παγκόσμια οικονομία και στο ελεύθερο εμπόριο. Αλλά όταν μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας, δεν λαμβάνει την απαραίτητη σημασία η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά μέχρι το 2020. Εγώ είμαι επιφυλακτικός για περαιτέρω δεσμευτικού στόχους και σας ερωτώ τι έχει βελτιωθεί από την Κοπενχάγη και τι έχει επιδεινωθεί για μια παγκόσμια λύση μιλάμε. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά συγκεκριμένα το εμπόριο εκπομπών. Εδώ πέρα υπάρχει μια σειρά θεμάτων που θα πρέπει να κρυθούν αυτή τη στιγμή. Θα τα αναφέρω. Κατανομή, ε, υπολογισμός και διαδικασία, οι δυνατότητες, οι νέες εγκαταστάσεις, όλα αυτά ζητήματα που πρέπει να κινηθούν βεβαίως σε ένα πλαίσιο συνένεσης, αναφέρθηκε ήδη στην κριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσει ο στόχος του 2020. Οπότε το ερώτημα είναι πώς θα δείτε αυτά τα ανοιχτά ζητήματα στο εμπόριο κουμπών. Ε, ευχαριστώ. Εντάξει λοιπόν, Φτάσαμε στο τέλος των ερωτήσεων. Το λόγο έχει πλέον η Επίτροπος για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον με τον κύριο Τόμψον, ο οποίος ε, επισημαίνει αμέσως το βασικό ζήτημα. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε με την Κίνα. Θα απαντούσα ναι, ακόμα μπορούμε. Όμως θεωρώ ότι προχωρούν ταχύτερα από ότι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Όταν θα δούμε το επόμενο πενταετές πλάνο τους, θα δούμε αυξηνόμενους στόχους για βιομηχανική ένταση, άλλους στόχους για τις ανανεώσιμες. Σύμφωνα με αυτά που είπαν, για πρώτη φορά θα έχουμε στόχους και εκπομπών και θα έχουμε και ενεργειακούς φόρους κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχω χρόνο για μακροσκελή απάντηση. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχει απειλή. Αν δεν είμαστε φιλόδοξοι στην Ευρώπη μπορούμε να χάσουμε θέση εργασίας. Αυτό το έθεσε και ο κύριος Λάγκεν. Αν το κάνουμε με τρόπο... Ε, πράγματι προχωρούμε με έναν τρόπο μη ευφυή, αλλά λέω ότι μπορούμε να το κάνουμε τρόπο ευφυή, που μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και τις, να, να πετύχουμε τους στόχους της καινοτομίας. Και επίσης βεβαίως υπάρχει το θέμα ότι μπορούμε να χάσουμε θέσεις εργασίας αν, αν δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι, γιατί όταν θέτεις φιλόδοξους στόχους, τότε δίνεις μια όθηση στις επιχειρήσεις για την καινοτομία. Και θα έλεγα ότι ο βασικότερος στόχος της Ευρώπη τα επόμενα χρόνια είναι να πετύχουμε περισσότερη καινοτομία για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε, να αντιμετωπίσουμε το διεθνή ανταγωνισμό. Ένα παράδειγμα για το πόσο γρήγορα κινείται η Κίνα. Πριν από 10 χρόνια η Κίνα δεν είχε ούτε έναν κατασκευαστή αιωλικής ενέργειας. Τώρα έχουν τρεις ε, εταιρείε αιωλικής ενέργειας, τις ανάμεσα στις 10 καλύτερες και αυτή τη στιγμή έχουν το 50% της παγκόσμιας αγοράς αιωλικής ενέργειας. Από 0 σε 10 χρόνια, μέσα σε 10 χρόνια έφτασαν στο 50% της παγκόσμιας αγοράς αιωλικής ενέργειας. Κάτι μας λέει αυτό για το τι, πόσο κινδυνεύουμε στην Ευρώπη. Πολλοί λοιπόν οι λόγοι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με σοβαρότητα έχουν κάνει σοβαρές επενδύσεις μέσω των πακέτων ανάκαμψης και αυτή τη στιγμή ανακοινώνουν ότι δεκαπλασιάζουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της αποτελεσματικότητας ενέργειας. Δεκαπλασιάζουν για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Μετά, η χρήση. Μπορούσα επίσης να είμαι μακροσκελής, θα είμαι σύντομη. Στις 14 Οκτωβρίου, στη διάσκεψη περιβάλλοντος, οι, Υπουργοί Περιβάλλοντος συμφώνησαν ότι εξωτερικά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις η Ευρώπη θα προσπαθήσει να ξεφορτωθεί τα, πλεον, τις, ε, ε, ε, τα, πλεονάζοντα δικαιώματα. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ τεχνικές συζητήσεις. Όμως, στην ουσία πρόκειται για 11 δισεκατομμύρια τόνους ζεστού αέρα στην ουσία δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Και το 2013, αν δεν γίνει κάτι, αυτό θα ε, εξαλείψει όλες τις πρωτοβουλίες της Ευρώπης μέχρι το 3%. Και θα, προσπαθήσουμε διεθνώς και στην Κανκούν να τα ξεφορτωθούμε. Και μετά θα δούμε πώς θα λύσουμε εσωτερικά το πρόβλημα. Και όπως υπηρετούμε σωστά, θα υπάρξει μια σωστή, ένας σωστός υπολογισμός του πακέτου αυτού. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η συζήτηση. Υπάρχει ένας εξωτερικός παράγων εδώ. Πρέπει αυτά τα επιπλέον δικαιώματα να τα καταργήσουμε. Ιδάλλως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές τους εσωτερικά. Ο Κλωτ Τούρμς με ρώτησε για την ανταγωνιστικότητα και το 30%. Όπως είπα, Πράγματι πιστεύω ότι αν προχωρήσουμε με έξυπνο τρόπο, πράγματι μπορούμε να ενισχύσουμε την καινοτομία. Αλλά έχει σημασία το πώς θα το κάνουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι εδώ ε, υπαναχωρούμε. Η ανακοίνωση του Μαΐου μας δείχνει ότι η Ευρώπη επιμένει στις υποσχέσεις που έδωσε διεθνώς. Αυτό είναι ένα σκέλος της ανακοίνωσης και το άλλο σκέλος αφορούσε το ότι για πρώτη φορά η Ευρώπη θα παρουσιάσει και ένα οικονομικό και βιομηχανικό συμφέρον. Έχει λόγους να είναι φιλόδοξη. Εμείς πιέζουμε και προχωρούμε σε αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε την Άνοιξη. Ο κύριος Σεντόμ με ρώτησε πώς θα πείσουμε ότι δεν είναι και τόσο κακό πλέον να είναι κανείς φιλόδοξος. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο σύμμαχο, τη βιομηχανία. Όλο και περισσότεροι κλάδοι συνειδητοποιούν, όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στην Κορέα και στην Βραζιλία, ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην εφησυχάζουμε. Αυτό βλέπουμε. Ένα παράδειγμα, στη συνάντηση των G20, την Πέμπτη. Ολόκληρη μέρα θα συναντηθούν τα στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο που θα ασχολούνται με την πράσινη ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι που πριν από μερικά χρόνια δεν θα συνέβαινε ποτέ. Επίσης, με ρωτήσατε για τη διαφάνεια για τη χρηματοδότηση. Θα πω απλώ ότι ναι, θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Στην Κανκούν η Ευρώπη θα παρουσιάσει επακριβώς το τι θα κάνει τι, ποιος θα κάνει τι. Θα αποδειχθεί ότι τα χρήματα θα παραδοθούν η απάντηση δεν είναι, είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι για όλα αυτά. Είδα τα ποσά από τα κράτη-μέλη και είπαν ότι δεν, δεν προστίθενται αυτά το ένα στο άλλο κατά 100%. Πρέπει όμως να πω ότι από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες να τους λέμε ειλικρινά τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, αντί να τους λέμε ότι αυτά είναι 100% επιπλέον ποσά, ενώ στην ουσία δεν είναι. Ο κύριος Οντί ρώτησε για τη διαδικασία του ΟΗΕ. Η εντύπωσή μου είναι ότι είναι δύσκολο, ρωτήσατε, ότι είναι δύσκολη διαδικασία. Η απάντηση είναι ναι, σαφέστατα. Ρωτήσατε αν μπορούμε να κάνουμε διμερεί ε, συμφωνίε. Ναι, ένα, ένα είναι αυτό το κάνουμε με την Κίνα, την Ινδία κλπ. Είπατε μπορούμε να πετύχουμε κάτι με την ε, Λατινική Αμερική, Μερκοσούρα α πούμε. Ναι, αν πρόκειται να κάνουμε μια εμπορική συμφωνία με τη Μερκοσούρ, τότε θα ενταχθεί σε αυτή και το περιβάλλον. Αυτό είναι ένα κομμάτι της προσπάθειάς μας. Αλλά θέλω να πω ότι ταυτόχρονα με όλα αυτά πιστεύω ότι μας συμφέρει, συμφέρει σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προσπαθούν να, επιδιώχουν, να πετύχουν μια συμφωνία σε επίπεδο ΗΠΑ. Όλοι βλέπουμε τις δυσκολίες του, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να, λέμε, να πούμε ποια είναι η εναλλακτική, όπου όλοι θα βρίσκονται σε ίση θέση. Ήδη νομίζω απάντησα την ε, ερώτησή σας για τη χρηματοδότηση και τα 2,4 δις. Φέτος θα τα δώσουμε και θα παραδώσουμε ε, μέχρι την Κανκούν πολύ περισσότερα για να ξέρουν όλοι. Τώρα για τα CDM. Έχετε απόλυτα δίκιο. Γίνονται στρεβλώσεις στο σύστημα. Και όπως ε, ξέρετε έχει κάνει μια ανάλυση η Κομισιόν για το NH3 και τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πολλά διακυβεύονται. Καθώς δίνουμε χρήματα στην Ινδία και την Κίνα. Αλλά τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Τους δίνουμε ένα περίεργο κίνητρο να συνεχίσουν να παράγουν το HFC 22 που παράγει κατόπιν το 23 γιατί κερδίζουν. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος τον οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σπάσουμε και γι' αυτό θα ζητήσω προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εν γέννη πρέπει να αναμορφωθεί το σύστημα CDM. Πράγματι, από τα 2.500 ε, έργα CDM το 95 πηγαίνει σε πέντε πολύ γνωστές ανεπτυσσόμενες χώρες. Μόνο 52 έργα από τα 2.500 πάνε στην Αφρική. 17 στην Νότια Αφρική, οπότε μόνο 35 έργα έχουν πάει συνολικά στην Αφρική. Είναι προφανές ότι το σύστημα πρέπει να αναμορφωθεί με έναν τρόπο ώστε να είναι περισσότερη κλαδική συνεργασία με τις αναδυόμενες οικονομίες και κατόπιν να εξυγχρονίσουμε και να απλωστεύσουμε τον συνήθι μηχανισμό CDM για να είναι καλύτερες οι επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αναφερθήκατε στο 30%. Είπα ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις, η Γαλλία, η Γερμανία, η Φιλανδία ε, ίσως όχι 30 αλλά 25%. Ε, ο, ο Δανός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30%. Εγώ νομίζω ότι κάποιες νέες χώρες κατανοούν ότι έχουν τεράστιο ενεργειακό δυναμικό. Και καταλαβαίνουν ότι αν χρησιμοποιήσει κανείς σωστά την ενεργειακή αυτάρκεια, τότε μπορεί να δημιουργήσει επιτόπου πολλές θέσεις ε, εργασίας ε, και επομένως απλώς πρέπει να δώσουμε κάποια ε, δυνατότητα μέσω του προπολογισμού να γίνει πιο ελκυστική αυτό, αυτή η δυνατότητα, αυτό το ενδεχόμενο να γίνει πιο ελκυστικό. Αναφερθήκατε σε ορθολογικούς στόχους για την Κανκούνα και ενδεχομένω εδώ υπήρξε μία παρανόηση. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε ε, ε, τόκους. Είπα απλώς ότι θα πρέπει πρώτα να δούμε ναι μεν τους στόχους ε, για το 2050 είπα απλώς ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο ενδιάμεσο ανάμεσα από το 2020 και το 2050. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εστιάζουμε για το τι θα γίνει το 2020. Ας πούμε, ε, στη, στον τομέα των ε, μεταφορών είναι πολύ καλό να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος που έχουμε για το 2030 ή και αργότερα ή ε, για την ενέργεια το ίδιο και νομίζω ότι και η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις γενικότερα ε, θα μπορούσαν πολύ καλύτερα να προβλέψουν τις κινήσεις τους εάν ήξεραν τι θα συμβεί και λίγο αργότερα. Μπορώ να προσθέσω αυτό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, στη συμφωνία της ε, Κοπεγχάγης έθεσαν στόχο για το 2025 και για το 2030. Έχουν λοιπόν κάποιους ενδεικτικούς στόχους. Ε, παρέμβαση Γκρίτς από την Πολωνία. Ναι, βεβαίως ε, καταλαβαίνω ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά μόνοι τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, γίνεται προσπάθεια επίτευξης διεθνούς συμφωνίας. Να σας πω όμως... Μερικές φορές όταν η Ευρώπη βγαίνει πολύ μπροστά δεν ε, κερδίζει ε, απαραίτητα. Πριν από μερικά χρόνια, δύο-τρία χρόνια, είμαστε οι μόνοι που είχαμε βάλει στόχους όσον αφορά την, ε, το κλίμα. Στη Κοπενχάγη όμως και η Ιαπωνία και η Ρωσία ήρθαν με νέες προτάσεις. Και κάποιες μεγάλες χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία, στο τέλος ακόμα και η Κίνα, η Σιγκαπούρη, η Κορέα, η Ινδονησία, η Νότια Αφρική και άλλες πολλές ε, έθεσαν στόχους, ε, ε, εγχώριους στόχους και οι περισσότερες χώρες του G20 για πρώτη φορά έβαλαν τέτοιους στόχους. Συμφωνώ βεβαίως ότι το θέμα του άνθρακα είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Ξέρω ότι πρέπει να ε, βελτιώσουμε την ε, κατάσταση. Ξέρω ότι πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα παγίδευσης αποθήκευσης. Τώρα, το φυσικό αέριο και η συγκριτική αξιολόγηση που αναφέρατε, βεβαίως εμείς θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε κάποιες ε, αρχές. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε, δεν έχουμε σύμφωνα με την οδηγία που πρέπει να ακολουθήσουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με άλλες μορφές ενέργειας. Ε, σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Λάγκε, ναι, βεβαίως δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Πιστεύω όμως ότι και η Ευρώπη έχει 30 ιστορία στον τομέα που καταδεικνύει ότι βάζοντας ε, πρότυπα ε, ε, τελικά παίρνοντας κάποιες σημαντικές έτσι, θέσεις, σιγά σιγά έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. που πούμε, φτάσαμε να έχουμε πιο καθαρά αυτοκίνητα από άλλους. Η οικονομία με το περιβάλλον θα πρέπει οπωσδήποτε να βρουν ένα ευφύ τρόπο έτσι ώστε να εργαστούν από κοινού με καλά αποτελέσματα. Γιατί διαφορετικά όντως μπορεί να είναι αντίθετες ιδέες σχετικά με την Κοπενχάγη. Πολλές είναι οι χώρες οι οποίες συνειδητοποιούν ότι εάν δεν δώσουμε συγκεκριμένα σημάδια προόδου στην Κανκούν, τότε κινδυνεύει η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών όχι να πεθάνει ακριβώς, αλλά ότι στην ουσία δεν θα έχει κανείς συμφέρον να την συνεχίσει. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι στο Μεξικό μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολλές οι χώρες οι οποίες θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν έτσι ώστε να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα κοιτάξτε, μέχρι τώρα η, η Ινδία και η Κίνα έχουν αρνηθεί να συζητήσουν το θέμα του κλίματος στην, ε, ε, στο G20. Το G8 το να το συζητάει δεν έχει και πάρα πολύ έννοια μεταξύ μας να τα λέμε. Ε, και επομένως νομίζω ότι πλέον έχουν όλοι αναγνωρίσει ότι είναι προς το συμφέρον όλων να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Τώρα θα σταθούν από επιτυχία, θα πετύχουμε, δεν το ξέρω, ειλικρινά σας λέω δεν το ξέρω. Νομίζω πάντως ότι κάτι που έχει ενδυναμωθεί από την ε, ε Κοπενχάγη είναι ότι οι επιχειρήσεις καταλαβαίνουν τι κάνουμε, η βιομηχανία καταλαβαίνει τι κάνουμε και ε, οι επιχειρήσεις θέλουν ένα κοινό ε, παρονομαστή. Δεν θέλουν 500 διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά κυρία Επίτροπε. Σας είμαστε ευγνώμονες που ήρθατε σήμερα εδώ ε, στην Επιτροπή μας για να μας πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν ναι, και αρκετά ενδιαφέρουσα και η ανταλλαγή των απόψεων νομίζω και πολύ ειλικρινής ε, κατά την άποψή μου. Και ξέρετε, και σας το λέω ειλικρινά, πολύ σπάνια παίρνουμε τόσο συγκεκριμένες απαντήσεις ε, σε συγκεκριμένες ερωτήσεις από τους ε, επιτρόπους. Γι' αυτό, εξ ονόματος των συναδέλφων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ πολύ δύναμη για τη συνέχεια των διπλωματικών σας διαπραγματεύσεων. Γεια σας.